και κατάργηση της οδηγίας 2004-8 και 2006-32. Έχουμε δύο στοιχεία σε αυτό το σημείο της ημέρησιας διάταξης. Καταρχήν μια συζήτηση για την έκθεση αντικτύπου και για τα ερωτήματα τα οποία θέσαμε σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Θα ήθελα εδώ να χαιρετήσω τον αρμόδιο επικεφαλής τμήματος και το δεύτερο τμήμα είναι η καλύτερη διευκρίνηση των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ένταση εργασίας, ενέργειας συγγνώμη, και έχουμε προσκαλέσει δύο εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα μας δώσουν τα φώτα τους σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αν συμφωνείτε λοιπόν, θα ήθελα να δώσω το, το λόγο σε ένα από τους καλεσμένους μας, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την συζήτηση και μετά να υπάρξει δυνατότητα να τεθούν και ερωτήματα. Έχετε λοιπόν τον λόγο, στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, όχι στους καλεσμένους. Θα δώσω το λόγο πρώτα. Σας ευχαριστώ. Δεν πρέπει να επανέλθουμε στα θέματα αυτά, αφού θέλουμε να μιλήσουμε για την έκθεση αντικτύπου. Μπορώ να σας συνοψίσω τα αποτελέσματα που, στα οποία καταλήγει η έκθεση αντικτύπου. Εξετάζουμε ένα αριθμό μέτρα για να κλείσουμε το χάσμα το οποίο υπάρχει μεταξύ της τωρινής πορείας και αυτού που είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους της Ευρώπης 2020 για την ενεργειακή απόδοση. Επί τη βάση λοιπόν αυτών των κριτηρίων εντοπίζουμε και ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνονται στην προτινόμενη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε η δική μας εκτίμηση για αυτά τα μέτρα είναι ναι, θα μας φέρουν στο στόχο του 20%. Δεύτερον, σε οικονομικούς όρους θα είναι θετική. Θα οδηγήσουν λοιπόν σε καθαρή αύξηση σε απασχόληση, 400.000 θέσεις απασχόληση και καθαρή αύξηση ΑΕΠ, 34 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020 και ένα μεγάλο μέρος αυτού του κέρδους θα είναι το γεγονός ότι αντικαθιστούμε εισαγόμενες πηγές ενέργειας με εγχώριες πηγές ενέργειας. Τρίτον, η πρόταση αυτή μαζί με τους στόχους του 20% για εξοικονομήσεις σε εκπομπές αερίων των θερμοκηπίων και αύξηση της αποδοτικότητας θα αύξαναν και το επίπεδο εξοικονομήσεων στα αέρια θερμοκηπίου. Δεν θα ήταν απλώς ένας διαφορετικός τρόπος για να επιτύχουμε το στόχο των αερίων θερμοκηπίου, αλλά δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα δεν μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα σαφές συμπέρασμα για το πώ θα έπρεπε να καταλήξουμε σε ένα τίμημα άνθρακο. Γι' αυτό η οδηγία προτείνει να το δούμε αυτό σε πιο πολλή λεπτομέρεια καθώ προχωρούμε την εξέταση των θεμάτων. Αυτό θα ήθελα να σταματήσω εδώ και είμαι έτοιμο να απαντήσω τα ερωτήματά σα. Μερσή λέει ο πρόεδρο. Έχει ξεκινήσει λοιπόν συζήτηση και θα ήθελα αυτοί οι οποίοι θέλουν να θέσουν ερωτήματα ενδεχομένω να το πράξουν. Ο κύριος Πίπα. Έχω την ευκαιρία μετά να επανέλθω. Κοιτάξτε, εγώ ε, θεωρώ εξυπνότερο να μην ρωτήσετε τώρα και να επανέλθω μετά. Ευχαριστώ. Α, εντάξει, τόσο ή δεν γίνεται και χαμός. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ρωτάω γιατί ακούστηκαν πράγματα που αφορούν το ερώτημα τη Κομισιόν. Καταρχήν ευχαριστούμε για το ότι απαντήσατε στα ερωτήματά μας τόσο γρήγορα. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν βεβαίως με ένα βασικό ερώτημα το οποίο θέλω να ξεκινήσω. Ξέρουμε πως το Συμβούλιο αρνείται να θέσει δεσμευτικό στόχο γιατί ακριβώς ορίζεται και ως στόχος εξοικονόμησης. Γι' αυτό σας ρωτήσαμε μήπως θα ήταν λογικότερο ως ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσετε, να ορίσετε αυτό το θέμα στην σχετική οδηγία και προσπαθήσαμε και εμείς να συνεισφέρουμε κάπως με τον εξή τρόπο να μην ορίσουμε μόνο τον απόλυτο στόχο εξοικονόμησης για το ισοδύναμο δηλαδή 380.000 τόνων πετρελαίου το οποίο είναι κάτι το αποδεκτό, αλλά προσπαθήσαμε να προτείνουμε και έναν τρόπο με τον οποίο μέσω υψηλότερης παραγωγικότητας της ενέργειας θα πάμε σε 104 τόνους ανά ε, εκατομμύριο ΑΕΠ. Και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σχετικός στόχος ε, ενέργειας ε, στον εξοικονόμηση που όλοι θέλουμε και τώρα μας κατηγορούν και δεν λάβαμε απάντηση ούτε από την Κομισιόν. Το ποιο θα ήταν το επιχείρημα που θα μπορούσαμε να φέρουμε όσον αφορά τη βιομηχανία με τον στόχο αυτό γιατί λέμε πως ε, δίνουμε προνόμια σε κάποιους κλάδους παρα... Ε, της ε, ενέργειας, γιατί λέμε δεν θέλουμε μόνο απόλυτο στόχο εξοικονόμησης, αλλά και μια σχετική μείωση της έντασης ενέργειας. Και ούτε η Κομισιόν μέχρι στιγμής δεν έχει δηλώσει γιατί με τον σχετικό αυτό στόχο εξοικονόμησης γινόμαστε πιο ελαστικοί σε σχέση με τον απόλυτο στόχο που είχαμε ορίσει τα 380. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Ε, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ή να αφήσω να απαντηθεί πρώτα. Παρακαλώ, έχετε λοιπόν την ευκαιρία να απαντήσετε αμέσως. Ευχαριστώ κύριε Πίπερ. Στην αξιολόγηση αντικτύπου αξιολογούμε τρόπους για το πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο του 20% όπως όρισε το 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και αυτό ορίζεται ως εξοικονόμηση 20% της κατανάλωσης σε σύγκριση με μια συγκεκριμένη προβολή και γι' αυτό το θέμα του ε, που ε, πηγαίναμε δεν το εξετάσαμε γιατί βεβαίως θεωρήσαμε πως ήταν κάτι το σαφές. Αντιλαμβάνομαι πως το ερώτημα του εάν αυτός ο στόχος θα πρέπει να επανεκφραστεί ως ένας στόχος έντασης ενέργειας είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει εντωμεταξύ στην πολιτική συζήτηση και αντιλαμβάνω πως είναι το αντικείμενο της συζήτησης με τους ειδικού και που θα ακολουθήσει. Εάν είναι να σας πω την άποψή μου, είναι πως η πρόταση της Κομισιόν είναι αυτή που είναι. Την έχετε δει, δεν εκφράζεται με αυτούς τους όρους, δεν έχουμε αλλάξει επισήμως. Δεν έχουμε μεταβάλει άποψη βεβαίω, ε, όπως και οποιοδήποτε άλλο θα ε, επανεξετάσουμε τη θέση μας για να δούμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε επικοδομητικά συμπεριλαμβανομένων και ιδεών που αφορούν την ένταση τη ενέργεια. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή στι θέσει κομισιών Μάρκος Πίπερ. Μάρκος Πίπερ. Ε, μου είπατε την ίδια αυτό που σας ρώτησα. Γιατί ο σχετικός στόχος δεν οδηγεί στο αποτέλεσμα 368 εκατομμύρια τόνους, όπως μας λένε πολλοί. Έχετε συγκεκριμένα δεδομένα. Μπορείτε να μας πείτε πως με τον σχετικό στόχο δεν θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Where you end up with. Το που θα καταλήξουμε με έναν σχετικό στόχο εξαρτάται από δύο πράγματα. Το πρώτον είναι σε ποιο επίπεδο ορίζουμε το στόχο και το δεύτερο είναι σε ποιο επίπεδο θα καταλήξει το ΑΕΠ να είναι και η κατανάλωση της ενέργειας. Οπότε δεν μπορούμε να αυτομάτως τι νούμερο θα δώσει ένα σχετικό στόχος, γιατί εξαρτάται και από τη φιλοδοξία του στόχου και στο τι συμβαίνει στο ΑΕΠ, οπότε δεν μπορεί να υπάρξει μια απλή απάντηση. Κυρία Χολ. Θα ήταν σωστό να πει κανείς με διαφορετικό τρόπο ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως έχει μπορεί να οδηγήσει στο, στη μείωση κατά 20% αλλά οι στόχοι έντασης της ενέργειας δεν θα πετύχουν τον συγκεκριμένο στόχο. Και γι' αυτό δεν έχουμε ακριβώς και μια τέτοια στοχοθεσία θα έλεγα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή δεν είναι μια συζήτηση που έχει και πολύ σχέση με τη μελέτη των επιπτώσεων, έτσι δεν είναι. στόχος της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να κάνουμε μια πρόταση επί τη βάση συγκεκριμένης αναλύσεως και σύμφωνα με την ανάλυση αυτή δεν θα πετύχουμε το 20%. Σας είπα πώς εμείς κατανοούμε το 20% στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Είναι μια μορφή εξοικονόμησης ενέργειας σχετικής με τις προβολές που κάνουμε εμείς. Είναι ένας αριθμός και όχι ένας στόχος έντασης ή χρήσης έντασης. Κάποιος άλλος. Α, ναι, Κλοντ Τούρμας. Of course I could add... Uh, μπορούσα να προσθέσω και εγώ κάποιες ερωτήσεις στην αξιολόγηση αντικτύπου, αλλά το ερώτημά μου απευθύνεται και προς τον κύριο Πίπερ και δεν ξέρω ποιος άλλος υπέβαλε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Εάν δεν έχετε νέες ερωτήσεις προς τις απαντήσεις της Κομισιόν. Μπορούμε να υποθέσουμε άρα πως η αξιολόγηση αντικτύπου και οι ερωτοαποκρίσεις, οι εκτεταμένες που προηγήθησαν μπορούν να σας κάνουν να θεωρήσετε πως η βάση επί της οποίας βασίζεται αυτή η οδηγία, δηλαδή η αξιολόγηση αντικτύπου, ότι δηλαδή δεν είμαστε στη σωστή πορεία, ότι έχουμε κάποιες προτάσεις, ότι οι περισσότερες από αυτές τις προτάσεις θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη ε, της Ευρώπης και σε θέσεις εργασίας, πως ε, υπάρχει άρα μία ευρεία συνένεση της Επιτροπής επ' αυτού και μπορείτε να το δεχτούμε ως βάση για τη συζήτηση μας. Το ερώτημά σας μπορεί να απαντηθεί βεβαίως όχι από την Κομισιόν, αλλά από αυτούς τους οποίους το απευθύνεται. Κοιτάξτε, για μένα προσωπικά δεν είναι και οι ερωτήσεις ε, ικανοποιητικές. Και εγώ το διάβασα και ε, μου δημιουργήθηκαν περισσότερα ερωτήματα από αυτά τα οποία απαντήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Φόρντ. Ευχαριστώ για το ίδιο θέμα και μένω στους αριθμούς που έχετε δώσει. Πολύ σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έδωσε κάποια στοιχεία αριθμητικά στα πλαίσια των αιτιολογικών σκέψεων ουσιαστικά για να δούμε ποια είναι η ένταση της ενέργειας στην γεωργία, στην βιομηχανία συγγνώμη, με τις εξοικονομήσεις στον τομέα της ενέργειας στους υπόλοιπους τομείς της δραστηριότητας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν καταλαβαίνω καλά, το κομμάτι που δεν ανήκει, εν πάση περιπτώσει, στη βιομηχανία, είναι το 269. Με, με απλή αριθμητική μιλάμε περίπου για τα 3 τέταρτα της μη βιομηχανική χρήσης της ενέργειας. Συμφωνεί και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, οπότε τρία τέταρτα του τομέα δηλαδή, ο οποίος μας απασχολεί, είναι από το 269, είναι το 269, συν κάποια μέτρα τα οποία αφορούν συγκεκριμένα τη βιομηχανία μπορείτε να καταλήξετε στην ίδια λύση. Η βιομηχανία έχει κάποιες ανησυχίες σε σχέση με τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να μας επιβεβαιώσει ότι οι αριθμοί τους οποίους έχω υποβάλει ή μας έχουν υποβάλει είναι σωστή έτσι ώστε η συζήτηση την οποία κάνουμε να είναι συζήτηση που να βασίζεται σε αυτά τα οποία πράγματι πρέπει να ξέρουμε. Παρακαλώ. Ε, ζητώ συγγνώμη, δεν έχω διαβάσει ακόμα τις αιτιολογικές σας σκέψεις. Οπωσδήποτε το νούμερο το οποίο αναφέρατε κάτι μας λέει είναι νομίζω 73% αντί για 75% στον ε, κλάδο. Μία ερώτηση σημαντική πολύ για μένα. Πώς μπορεί κανείς να καθορίζει στόχους εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς να κάνει την αντιστοίχηση με τις πραγματικές ανάγκες και με τις προσπάθειες να ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτές. Υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία ακούγονται θα ασχοληθώ με ένα. Ας φανταστούμε, δικαιωμά μου ας είναι, ότι εν τη πλήρη αυτή σοφία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει ότι θα πρέπει να επιταχύνει τη βιομηχανική δραστηριότητα, να παράγονται όλο και περισσότερο προϊόντα σε τοπικό επίπεδο για να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, σαν παράδειγμα για να εξοικονομηθεί διοξίδιο του άνθρακα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στο σιδηροδρομικό τομέα έτσι ώστε τα εμπορεύματα να μετακινούνται με τρένο ή επιβάτες να μετακινούνται με τρένο σε όλα τα μέρη της Ευρώπης. Ας τα φανταστούμε όλα αυτά. Ας φανταστούμε επίσης ότι ο ευρωπαϊκός πληθυσμός συνεχίζει να εξελίσσεται όπως σήμερα. Το ερώτημα το οποίο τίθεται λοιπόν είναι ότι πριν ξεκινήσει να κάνει εξοικονόμηση ενέργειας η Ευρώπη είναι σε θέση να παράγει την ενέργεια την οποία χρειάζεται. Δεν ξέρω. και μεγάλη σχέση βέβαια με την... Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σχέση το ερώτημα αυτό με το ζήτημα της σε αντικτύπου. Μα ο, αναφέρθηκε και σε μένα ο Κλοντ ε, Τούρμες. Ε, ζητώ συγγνώμη, ήταν η πρώτη ερώτηση, είπα πως είχα και άλλες ερωτήσεις, δεν έχουμε ολοκληρώσει. Σε, με συγχωρείτε, θα ακολουθήσουν και άλλες. Θα ήθελα να έρθω στο ερώτημα 4, στην κοινή μέθοδο μέτρησης. Γράφεται πως η πρόταση δεν έχει κοινή μέθοδο μέτρησης για την εξοικονόμηση ενέργειας και τα σχετικά μέτρα. Θα αναφέρω μία μελέτη του Ινστιτούτου Φράουνχόφερ. Να αναφέρομαι τώρα στο άρθρο 6 της πρώτας οδηγίας. Εάν σε τέσσερις χώρες, Δανία, Ιταλία, Βέλγιο και Γαλλία, αλλάξουμε τα ψυγεία, ε, οδηγόμαστε σε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα εξοικονόμησης σε αυτές τις τέσσερις χώρες. Υποθέτει η Κομισιόν πως κάθε χώρα θα μετράει διαφορετικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίπερ, στην απάντησή μας στην ερώτηση 4 είπαμε πως δεν προτείνουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πολύπλοκες ε, μεθόδους ε, μέτρησης που προσπαθούμε να αναπτύξουμε υπό την υφιστάμενη οδηγία ε, υπηρεσιών ενέργειας και προτιμούμε να πάμε όχι σε μη μέθοδο μέτρησης αλλά σε μία απλούστερη. Και το πρόβλημα ήταν βεβαίως πως δεν υπήρχε συνένεση μεταξύ των κρατών μελών για το πώς θα πρέπει να γίνει αυτό. Για τη μελέτη του Ινστιτούτου Φράουνχόφερ έχω διαβάσει μια σύνοψη και όχι ολόκληρη τη μελέτη, αλλά το συμπέρασμα που αναφέρεται είναι απολύτως σωστό. Εάν δείτε τη... τα συστήματα υποχρέωσης ενεργειακής αποτελεσματικότητας, βλέπουν το ίδιο μέτρο με τελείω διαφορετικό τρόπο όσον αφορά το αποτέλεσμα, το όφελο που έχει. Δεν θέμε αυτό το αποτέλεσμα παρά το ότι βεβαίως στόχο έχουμε να έχουμε μία ενιαία εναρμονισμένη ευρωπαϊκή μέθοδο μέτρησης, αλλά στο παράδειγμα 5 ορίζουμε κάποιες βασικές κοινέ μεθόδους μέτρησης, Έλεγε πως εάν τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν άλλη μέθοδο, πρέπει αυτή να κοινοποιηθεί στην Κομισιόν και η Κομισιόν θα έχει τη δυνατότητα να δει εάν είναι τουλάχιστον το ίδιο φιλόδοξη με αυτά που αναφέρει η οδηγία. Ευχαριστώ.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 την δυνατότητα εξοικονόμησης και μιλάτε για τους 368 ε, εκατομμύρια τόνους κτλ. Θα αναφέρω κάποια παραδείγματα στην αξιολόγηση αντικτύπου για το 2011. Αναφέρεται πως μόνο τα 11 μέτρα που έχουν αποφασιστεί για τον οικολογικό σχεδιασμό ε, σημαίνουν 83.000 ε, τόνους οικονομία μέχρι το 2020. Μα υπάρχει και άλλο ένα μέτρο στο eco-design Οπότε πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα. Τώρα, για την ε, συλλογική, συνολική αποτελεσματικότητα των κτηρίων. Η Κομισιόν διαπιστώνει πως τα μέτρα τα οποία προτείνονται εκεί σημαίνουν 96 εκατομμύρια τόνους εξοικονόμηση, δυνατότητα εξοικονόμησης. Οπότε έχουμε φτάσει 79 εκατομμύρια τόνους και λέτε μετά με ένα συντηρητικό υπολογισμό των προτινόμενων μέτρων μιλάμε για 107 ε, εκατομμύρια τόνους. Και συντηρητικό σημαίνει πως αυτό είναι το μήνυμο. Μήπως υπάρχει ο κίνδυνος ε, να εξοικονομήσουμε περισσότερο από όσο θα θέλαμε. Καλό θα ήταν. Ή δεν καταλαβαίνω, εν πάση περιπτώσει, τα μαθηματικά σας εδώ πέρα. Σε άλλα στοιχεία υπάρχουν αλλού νούμερα και ξαφνικά το σύνολο είναι μεγαλύτερο. Δεν, δεν μου φαίνονται πολύ κατανοητά αυτά. Μετά, στην ερώτηση 36, το ποια περαιτέρω εμπόδια μπορούν να υπάρξουν σε αυτόν τον τομέα. Ποια είναι τα εμπόδια τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσει το εμπόριο εκπομπών για την περαιτέρω επέκταση αυτού του συστήματος. Ε, πείτε μας, δηλαδή, ποια, είναι τα, τα εμπόδια. Αυτές τις ερωτήσεις θα ήθελα εγώ. Θα μπορούσατε να απαντήσετε. Τα κέρδη από τα προγράμματά μας και συγκεκριμένα η επέκταση της οδηγίας για την οικολογική σχεδίαση σε προϊόντα τα οποία ε, εμπλέκονται στην εξοικονόμηση ενέργειας, η αξιολόγησή μας βασίζεται στο βασικό σενάριο, δηλαδή ότι χωρίς καμία απολύτως δράση μπορούμε μέχρι το 2020 να πετύχουμε μια εξοικονόμηση 10%. Έχουμε τώρα προσθέσει εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο αυτών των μέτρων. Μια μεγάλη δυσκολία. Με οποιαδήποτε αξιολόγηση για τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας είναι ότι αυτά τα μέτρα επικαλύπτονται και ενισχύουν τα μέντα, δε και δεν είναι καθαρά προσθετικά. Παράδειγμα, ένας από τους καλύτερους τρόπους να πετύχουμε τους στόχους της οδηγίας για τα κτίρια είναι να χρησιμοποιήσουμε καλύτερο κλιματισμό, καλύτερους λέβητες, καλύτερο φωτισμό. Και επομένως με το να υπάρχει κάποιο κίνητρο για τα ε, υλικά αυτά, δίδεται το κίνητρο. Από την άλλη μεριά η οδηγία για τις οικολογικές ε, ετικέτες ουσιαστικά εξαλείφει τα λιγότερο ενεργειακά ε, αποδοτικά από αυτά τα από το φωτισμό, τους λέβητες κτλ. Έχετε δει λοιπόν δύο ενέργειες οι οποίες ε, λειτουργούν παράλληλα αλλά δεν έχουν προσθετικά αποτελέσματα. Ζητήσαμε από τους υποδειγματίες μας αυτούς οι οποίοι κάνουν μοντέλα να είναι προσεκτικοί για να μην υπερτιμήσουν τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών και μετά από πολλές προσπάθειες σε σχέση με τα μέτρα αυτά και τις μελέτες μας καταλήγουμε στα στοιχεία που έχουμε στην έκθεση αντικτύπου. Τα μέτρα λοιπόν αυτά που προτείνουμε όπως είναι η, η υποχρέωση για ανεργειακή απόδοση θα δημιουργήσουν περαιτέρω εξοικονόμηση και επομένως αυτή η διπλή καταμέτρηση λαμβάνεται υπόψη για τη συμπαραγωγή ενέργειας και θερμότητος η... περιλαμβάνεται υπόψη η παραγωγή ηλεκτρισμού από τους ε, συνδυασμένους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και θερμότητας, δεν καταμετράται και <clears throat> ο αντίκτυπος της θερμότητας. Αυτό σημαίνει και μια έλλειψη επαρκών κινήτρων για το σύστημα αυτό συνδυασμένης παραγωγής. Γι' αυτό για μας το σύστημα εμπορίας εκπομπών δεν έχει επιτρέψει να εκμεταλλευτούμε πλήρως το δυναμικό αυτών των σταθμών. Ελπίζω ότι έτσι απαντώ στα ερωτήματά σας. Ο Μάρκους Πίπα. χωρίς μικρόφωνο. Θέλω να πω κάτι για το θέμα χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Λέτε εδώ πέρα πως πολλά από αυτά τα μέτρα, ειδικά για το δημόσιο τομέα, από το 2014 πιθανώς θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία. Εδώ πέρα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως ήδη στις σχετικά πλουσιότερες περιοχές, μιλάμε για ένα 50% τουλάχιστον συγχρηματοδότησης. Και τα χρήματα αυτά, τα πολύτιμα των διαρθρωτικών ταμείων πρέπει και υπάρχει ο ανταγωνισμός να καλύψουν ε, ευρυζωνικότητα, επικοινωνίες, ε, βιολογικά διάφορα. Δεν έχω ιδέα. Τέλο πάντων, διάφορα πράγματα μπορούν να απτύξουν μια περιφέρεια. Και θέλω να ρωτήσω πόσο σίγουροι μπορεί να είστε και θα υπολογίζετε αυτά τα χρήματα. Πώς ξέρετε πως οι περιφέρειες ε, έχουν τις ίδιες προτεραιότητες με εσάς. Εκτός εάν υπολογίζετε σε μια ε, νομοθετική υποχρέωση. Μήπως περιορίζεται δηλαδή τη χρήση των χρημάτων των διαρθρωτικών ταμείων. Πρώτο ερώτημα. Άν μου επιτρέπετε άλλο ένα ερώτημα. Αναφέρθηκα επίσης στην απάντησή σας στο ερώτημα 7 τώρα να αναφερθώ στο ερώτημα 12. Ρωτήσαμε εδώ γιατί το 1,5% το ποστό εξοικονόμησης είναι το ίδιο σε όλες τις χώρες. για να επιτευχθεί ο στόχος του 20%. Αν υπάρχει κάποια αιτιολόγηση. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι η αφετηρία του κάθε κράτους μέλους διαφέρει πάρα πολύ. Και ρωτήσαμε γιατί αιτιολογείται αυτή η ίση αντιμετώπιση όλων των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Για το θέμα των διαφθορτικών ταμείων νομίζω ότι αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση. Εν μέρη μπορώ να απαντήσω. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύπτει περίπου 17 δις ευρώ μέσω των διαφορετικών για το πολιετές πλαίσιο 14-20 το οποίο θα πρέπει να προσημειωθούν κατά κάποιο τρόπο τα χρήματα αυτά για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτή είναι η πρόταση. Ποια θα είναι η τελική απόφαση ή θα το αποφασίσουν οι συνομοθέτες. Για το 1,5%. θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι κάτι το οποίο ρυθμίζεται σε θελοντική βάση και αυτό που έχει σημασία είναι η εθνική στόχοι. Και γι' αυτό ακριβώς, ορίζοντας τους στόχους αυτούς τα κράτη-μέλη, είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβουν υπόψη τους το δυναμικό το οποίο έχουν ανεκμετάλλευτο και τι δυνατότητες εξοικονόμησης περαιτέρω υπάρχουν. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας προτείνουμε να υπάρχει ένα μόνιμο 1,5% το οποίο να εξοικονομείται από τους καταναλωτές μέσω των παροχαίων ενέργειας. Ακόμα και οι χώρες λοιπόν που έχουν πετύχει την μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας τα προηγούμενα χρόνια, χώρες όπως η Δανία σαν παράδειγμα, είναι σε θέση να μας δώσουν αυτό το 1,5% επιπλέον. Και γι' αυτό δεν υποστηρίζουμε την άποψη ότι ακριβώς αυτές οι προληπτικές δράσεις θα αποτρέψουν κάποια κράτη-μέλη να κάνουν το κάτι περαιτέρω, το οποίο είναι δυνατό να γίνει. Αντίθετα πιστεύουμε ότι υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στα προληπτικά μέτρα ή στα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σε μια πρώιμη περίοδο και στα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σε τακτική ετήσια βάση. Ευχαριστώ και ένα ερώτημα εγώ να προσθέσω το οποίο το είχα ξεχάσει πριν. Στο θέμα 45, σημείο 45. Το ερώτημα είναι το εάν η Κομισιόν έκανε την ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους σε διαφορετικά σημεία και πόλεις και κατέληξε πάντα στο ίδιο συμπέρασμα και αναφέρεται ως παράδειγμα τη Βαρκελόνη. Με ενδιαφέρει, είχατε και άλλες πόλεις και ποιες. Και, ε, και άλλες πόλεις, αν ήταν μικρές πόλεις και ποιο ήταν το αποτέλεσμα γιατί βεβαίως μία χώρα, ξέρετε, με μικρότερες πόλεις ε, θα είχε διαφορετικά αποτελέσματα. Οπότε το ερώτημα είναι αν ε, είχατε και άλλες πόλεις και ποιες ήταν αυτές, εάν είχατε. These systems operate successfully in towns much smaller than Barcelona. However, um, I'm afraid that τα συστήματα αυτά λειτουργούν και σε μικρότερες αστικές συγκεντρώσεις από αυτή της Βαρκελόνης. Mm. αλλά δυστυχώ δεν έχω τις λεπτομέρειες τη μελέτη αυτή και γι' αυτό να μου επιτρέψετε να σας στείλω γραπτά τις λεπτομέρειες σχετικά με τις πόλεις στις οποίες υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Σας ρώτησα γιατί είπατε ότι στην απάντησή σας είπατε ότι είχατε κάνει χωριστές αναλύσεις στα θέματα αυτά ώστε να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος. Μήπως δεν μας πείτε για ποια μέρη κάνατε αυτή την, ε, για ποιες πόλεις, για ποιες τοποθεσίες κάνατε αυτή τη μελέτη, γιατί αλλιώς δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε. Για τα ευφύ κύτταρα, για, τα εφή, για τους εφείς μετρητές, συγγνώμη, αναφέρατε επίσης ότι υπάρχει μια σημαντική εξοικονόμηση Τι θα γινόταν κατά την άποψη της Κομισιόν αν είχαμε μια κάλυψη αντί για 50-70% στους ευφυείς μετρητές. Ποια θα ήταν η διαφορά λοιπόν, ποια θα ήταν η ψαλίδα η οποία θα μπορούσε να προκύψει αν δεν είχαμε μια πλήρη κάλυψη από τέτοιου μετρητές. Και η Κομισιόν άφησε επίσης ανοιχτό ένα ερώτημα για τις μελέτες που λένε ότι μόνο 40% των νοικοκυριών θα χρησιμοποιήσουν αυτούς τους ευθύς μετρητές, λέει αυτή η μελέτη. Ότι δεν θα είχε ε, επαρκή σχέση κόστους οφέλους για να τα, το, τους υιοθετήσουν όλα τα σπίτια και εδώ ήθελα να ξέρω αν η Κομισιόν σκέφτεται να έχει και περαιτέρω μέτρα για να προωθήσει την υιοθέτηση αυτών των μετρητών. Η αφετηρία μας είναι η νομοθεσία για την εσωτερική αγορά που ζητά από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν το ότι πράγματι είναι αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος να χρησιμοποιήσουμε ευφύης μετρητές για το φυσικό αέριο και για τον ηλεκτρισμό και στην περίπτωση του ηλεκτρισμού αν είναι πραγματι λογικό να φτάσουμε σε ένα 80% κάλυψης μέχρι το 2020. Τα κράτη-μέλη λοιπόν κάνουν αυτή τη στιγμή βάση αυτής τη νομοθεσία την εκτίμηση για τη σχεση κόστου κόστους-οφέλους αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σας πω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτών των μελετών. Για αυτό το λόγο και για άλλους λόγους δεν μπορώ να σας πω ποιο ποσοστό εφαρμογή των εφιών μετρητών μπορεί να επιτευχθεί. Τουλάχιστον θα έχουμε 50% μεγαλύτερο όφελος, αν είναι 50% 33% αν είναι μονάχα ένα τρίτο από αυτό το οποίο προστοκείται. Αν δεν έχουμε πλήρη κάλυψη θα έχουμε τουλάχιστον αναλογικά ωφέλη. Γιατί λέω τουλάχιστον αναλογικά, γιατί αν αυτό βασίζεται σε μια μελέτη κόστους-οφέλους, εκεί που δεν θα εφαρμοστούν οι μετρητές είναι γιατί έχουμε περιπτώσεις που υπάρχει λιγότερο, λιγότερο δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας και γι' αυτό δεν θα υπάρχει χρησιμοποίηση ευφυών μετρητών. Οι ευφυεί μετρητέ θα μπουν εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονόμηση. Δεύτερον, η πρότασή μα απαιτεί από του ε, καταναλωτέ να έχουν τακτικά πρόσβαση σε λογαριασμού ενέργεια, ακόμα και όταν δεν έχουν ευφυεί μετρητέ, με το να υπάρχει δυνατότητα να έχουν ένα σύστημα που να μπορούν να διαβάζουν μόνοι το λογαριασμό τους. Ακόμα και χωρίς ευφυείς μετρητές, σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να έχουμε κάποια εξοικονόμηση. Για αυτού τους λόγους ελπίζουμε ότι ακόμα και μια μερική χρησιμοποίηση εφιών μετρητών θα δώσει αποτέλεσμα το οποίο θα είναι υπεραναλογικό. Ωραία. Όσο δεν έχουμε τα στοιχεία των μελετών, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια συγκεκριμένη πρόβλεψη. Υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα από τους συναδέλφους. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος θέλει το λόγο. Έρχομαι στο θέμα των ερωτήσεων που έχουν να κάνουν με τους ελέγχους, τους απολογισμούς για τις ε, ενεργείες, ενεργείες τα λεγόμενα energy audits. Εάν δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις που να μπορούν να υποφελθούν από τέτοιους ελέγχους ενέργειας, τότε δεν πρέπει να υπάρχει και υποχρέωση για αυτούς. Η Κομισιόν λέει ότι πρέπει να βγουν από αυτό το, αυτήν την υποχρέωση η λογιστικού ελέγχου ενέργειας οι επιχειρήσεις που ήδη κάνουν κάποιο εσωτερικό έλεγχο για τις ενέργειες. Τι νόημα έχει αυτό που λέτε, ότι δεν χρειάζεται να γίνει έλεγχος επειδή αυτές ήδη τον κάνουν τον έλεγχο. Δηλαδή άμα τον κάνουν δεν πρέπει να τον κάνουν και άμα δεν τον κάνουν πρέπει να τον κάνουν. Πώς καταλήγει η Κομισιόν σε αυτή τη λογική και ποιο, εάν πρόκειται για μια εξαίρεση, ποιο θα επομιστεί το κόστος για κάτι τέτοια. Εγώ βλέπω να υπάρχει μια αντίφαση. Η πρότασή μα είναι μόνο μεγάλε εταιρείε να κάνουν τέτοιου ελέγχου κάθε τρία χρόνια και μικρέ εταιρείε δεν θα πρέπει να το κάνουν υποχρεωτικά. Αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν συστήματα που θα τις βοηθήσουν να έχουν ε, πρόσβαση στα ωφέλη των ενεργειακών ελέγχων. Η πρόταση αναγνωρίζει πως υπάρχουν ήδη ενεργειακοί έλεγχοι που γίνονται στο πλαίσιο εθελοντικών συμφωνιών ή συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και πώς αυτοί οι έλεγχοι, αν συμβαίνει αυτό, επαρκούν για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις ε, που προβλέπουμε. Οπότε δεν προβλέπουμε εξαιρέσεις στην υποχρέωση, απλά να αναγνωρίσουμε πως ήδη γίνεται ή κάτι τέτοιο εντός των υπαρχόντων συστημάτων. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Τίποτα άλλο από αυτό το μοντέλο. Γιατί το είχαμε συζητήσει και ήταν πολύ προβληματικό. Ακούω πως η Κομισιόν πλέον δεν είναι τόσο πολύ υπέρ αυτού του μοντέλου. Και μου είπαν πως τώρα είναι κάπως τα πράγματα κάπως υπάρχει μια βεβαιότητα. Τόσο. Θα ήθελα να γνωρίζω τι γίνεται εδώ πέρα. Νομίζω ότι μιλάτε. για το μοντέλο των ε, διαφόρων των Primes και έχουμε μία σύμβαση με αυτή την εταιρεία οπότε θα αναπτύξουν ε, το βασικό μοντέλο δηλαδή το τι θα συνέβαινε με το να συνεχίσουν τα πράγματα ως έχουν, γιατί όπως σας είπα εμείς λαμβάνουμε υπόψη τα μέτρα μέχρι το τέλος του 2009. Προετοιμάζουμε μία βεβαίως ενημέρωση που θα λαμβάνει υπόψη και το τέλος του 2011 με τους ειδικού ε, της στατιστικής. Βεβαίω δεν είναι αυτό μόνο, το μόνο μοντέλο που έχουμε και οπωσδήποτε θεωρούμε πως είναι αναγκαίο να κοιτάξουμε τα αποτελέσματα και σε σχέση με τα δικά μας μοντέλα και σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο Ινστιτούτο. Μάλιστα. Τώρα, δεν με ενδιαφέρει τη σύμβαση που έχετε με αυτούς τους ανθρώπους. Με ενδιαφέρει το μοντέλο. Αυτό νομίζω ήταν ερώτημα των συναδέλφων. Εάν το μοντέλο αυτό είναι σωστό. Δεν είναι ε, ασήμαντη αυτή η ερώτηση. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες για αυτό το μοντέλο, ε, πρέπει να ξανασκεφτούμε ορισμένα πραγματάκια. Και λέτε τώρα πως θα συμπεριλάβετε και άλλα μοντέλα. Αυτό για μένα είναι ένδειξη πως δεν είμαστε 100% σίγουροι ας πούμε και επίσημοι, να το πω έτσι προσεκτικά. Ναι, ναι, η κυρία Ντελκαστίγιο παρακαλώ. Ε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το μοντέλο αυτό όπως ε, μπορείτε να κατανοήσετε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε μια μεγάλη ανησυχία πρόσφατα σε σχέση με τις επικρίσεις και τα ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί για το υπόδειγμα αυτό από διάφορα μέσα ενημέρωσης. Κατά πόσο είναι έγκυρο δηλαδή αυτό το μοντέλο. Αυτό το οποίο λέγανε ήταν ότι υπάρχει μια έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με, τη μαθηματική βάση του μοντέλου και η, η αδυναμία να το διασταυρώσουμε με άλλες ε, μελέτες μας αναγκάζει να έχουμε μια τυφλή εμπιστοσύνη στη λειτουργία του μοντέλου και στις προβλέψεις του. Δεν ξέρω λοιπόν αν υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα, γιατί αν υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί έχουμε κάποιες ε, κάποια συμπεράσματα αυτού του μοντέλου που δεν μπορούμε να τα διασταυρώσουμε με άλλο τρόπο. Υπάρχει λοιπόν η ανησυχία μήπως είναι λανθασμένα αυτά τα συμπεράσματα. Η Κομισιόν τώρα ξέρει τι ακριβώς έχει αυτό το μοντέλο. Θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν το θέμα του τι περιέχει αυτό το μοντέλο. Αυτό ήταν και το ερώτημα του Πρόεδρου από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Κλοντ Τούρμας. για την ε, κατασκευή των μοντέλων και τις προσωμιώσεις. Εγώ θα ήθελα να ζητήσουμε τους αρμόδιους στην Κομισιόν, ο κύριος ή τον αρμόδιο στη διεύθυνση που ασχολείται με την κατασκευή σεναρίων που αντιμετωπίζουν και το θέμα αυτό γιατί και τα δικά του σενάρια οικοδομούνται από τη βάση αυτού του μοντέλου. Θα ήταν χρήσιμο κάποια μέρα να έχουμε μία συζήτηση όπου να μας εξηγήσουν τι είναι τα primes, τι είναι αυτά τα οποία ονομάζουν delivering και ποια είναι τα, οι προτάσεις και τα συμπέρασμα της Κομισιόν για το μέλλον. Αυτό όμως υπερβαίνει τη σημερινή συζήτηση για την αποδοτικότητα της ενέργειας. Currents. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το μοντέλο. Σε όλη τη συζήτηση χρησιμοποιούμε το μοντέλο Primes ως βάση. Θεωρούμε ότι χωρίς καμιά αλλαγή αυτό θα λάβει χώρα και αν επιτύχουμε κάποιους στόχους θα έχουμε μια βελτίωση της κατάστασης, ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Αλλά όπως είπε και η συνάδελφός μου, εγώ δεν ξέρω πώς λειτουργεί το μοντέλο Prime αυτό είναι το πρόβλημα. Φαίνεται ότι κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το μοντέλο. Είναι γεγονός, όπως είπαν τα μέσα ενημέρωσης, ότι είναι μονάχα μια μικρή ερμητικά κλειστή ομάδα ερευνητών που είναι σε θέση να ελέγξει τα αποτελέσματα αυτού του μοντέλου. Ξέρει η Κομισιόν αν έχει υπάρξει μια ανεξάρτητη επαλήθευση αυτού του μοντέλου του Πράνς. Είναι έγκυρο το μοντέλο αυτό γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι βασικό για τη συζήτησή μας. Αν υπάρχουν δημόσια εξε... εκφραστήσεις αμφιβολίες για το μοντέλο του οποίου εδράζεται η νομοθεσία μας, θα πρέπει να ξέρουμε κάτι περισσότερο. Θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η πιθανότητα αυτό το μοντέλο να είναι έγκυρο και πόσο να μην είναι έγκυρο. Μπορεί η Κομισιόν λοιπόν να καταπράγει τους φόβους οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί έχουν διατυπωθεί δημόσια σε σχέση με το μοντέλο αυτό που χρησιμοποιείται σαν βάση για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Ο κύριος Πίπα. Ευχαριστώ. Απορώ λίγο για το ότι ο κύριος Χότσον ομολογεί πως υπάρχουν και άλλα επιστημονικά μοντέλα. Και εμείς θα θέλαμε να έχουμε κάποια άλλη βάση. Τώρα, εάν η βάση του Πολυτεχνείου της Αθήνας ε, δεν ισχύει πλέον το μοντέλο, το πανεπιστήμιο το οποίο δημιούργησε αυτό το μοντέλο, ε, θα ήθελα να μας το κάνετε κάπως πιο συγκεκριμένο. Οπότε παρακαλώ να μας ξεκαθαρίσετε ε, πόσο πραγματικά αξιόπιστο είναι αυτό το μοντέλο. Έχετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα και ίσως είναι ε, το ευκολότερο αυτό να σας πω τι ρόλο παίζει το μοντέλο Primes σε αυτά τα οποία βλέπετε μπροστά σας. Ο βασικός ρόλος είναι πως έτυχε να είναι η προβολή η οποία υπήρχε το 2007 Οπότε ήταν η γλώσσα η οποία χρησιμοποιήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για να ορίσουν μια αφετηρία από την οποία μετά θα αφαιρούσαν ένα 20%. Ήταν δηλαδή μια συγκεκριμένη λειτουργία του μοντέλου Primes με, για να οριστεί ο στόχος 100. Και αυτό, γι' αυτό υπάρχει αναφορά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Αν δείτε τώρα τι άλλο ρόλο παίζει στην πρότασή μας, θα δείτε πως η απάντηση είναι πολύ λίγο. Αν δείτε την οδηγία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προτείνουμε δεσμευτικούς στόχους για τα κράτη-μέλη. Οι στόχοι αυτοί δεν βασίστηκαν στο ε, μοντέλο Prime ή οποιοδήποτε άλλο μοντέλο. Είδαμε που ήταν τα κράτη-μέλη και από εκεί προτείναμε. Και άρα δεν προτείναμε δεσμευτικούς ε, στόχους, αλλά προτείναμε άλλα νούμερα για στόχους, οπότε δεν βασιζόμαστε στο μοντέλο Prime σε αυτή την αξιολόγηση. Αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε, και έρχομαι στο ερώτημα του κυρίου Πίπερ, χρησιμοποιούμε το μοντέλο Primes μεταξύ άλλων για να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο των διαφόρων μέτρων που προτείνουμε. Ο κύριος Ρόιλ ρώτησε αν είμαστε 100% σίγουροι η απάντηση είναι 100% όχι. Όποιο μοντέλο και να έχουμε, όποια εταιρεία και να το κάνει, όσο διάφανη και να είναι η μέθοδος, οποιοδήποτε ε, ερχόταν και σας έλεγε ναι, θα σας κοροϊδεύε. Γιατί ε, εξορισμού τα μοντέλα είναι κάτι το αβέβαιο. Χρησιμοποιούμε το μοντέλο Primes και προσπαθούμε να συμφωνήσουμε τα κράτη-μέλη στι υποθέσει που βάζουμε σε αυτό, αλλά στην αξιολόγηση αντικτύπου, και εδώ πέρα έρχομαι σε αυτό το οποίο είπε ο κ. Πίπερ, χρησιμοποιήσαμε επίση το μοντέλο E3ME τη Cambridge Econometrics, μια εταιρεία όσον αφορά την αξιολόγηση των μέτρων μας. Κάποιες φορές ήταν στο ίδιο αποτέλεσμα, άλλες φορές όπως την τιμή του άνθρακα ήταν σε διαφορετικό, κατέληξε σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Τα λέμε όλα αυτά στην αξιολόγηση αντικτύπου επιπλέον. Όταν μιλάμε για συγκεκριμένους κλάδους, χρησιμοποιούμε μοντέλα που είναι σχεδιασμένα για αυτούς τους κλάδους. Οπότε, στα κτίρια έχουμε το μοντέλο BEAM και ούτω καθεξής. Αυτό πάντα συνέβαινε. Ε, δεν βλέπω εγώ εδώ πέρα κάποια παραχώρηση είναι απέτηση, αν θέλετε, της επαγγελματικής μας ευθύνη να αξιολογήσουμε από διαφορετικέ σκοπιές τον αντίκτυπο. I'm Ευχαρίστως να απαντάω σε ερωτήσεις για τον ρόλο του Prime σε σχέση με την πρόταση που έχετε τώρα μπροστά σας. Μπορώ επίσης να πω πως είναι μοιραία ένα ευρύτερο ερώτημα. Θα ήταν λάθος η Κομισιό να χρησιμοποιεί ένα μοντέλο σε μια πολιτική που έδινε καλά αποτελέσματα γι' αυτό και ένα άλλο μοντέλο διαφορετικό σε άλλη πολιτική. Λογικό είναι να χρησιμοποιούμε ένα ενιαίο μοντέλο σε όλες αυτές τις συζητήσεις. Οπότε μπορεί να γίνει πράγματι μια γενικότερη συζήτηση για το αν είναι σωστή αυτή η επιλογή για τα υπέρ και τα κατά. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι όλα τα μοντέλα που εξετάσαμε έχουν δυσκολία στο να δουν την πλευρά της ζήτησης από ότι σε ζητήματα προσφοράς. Ε, γιατί οι άνθρωποι βεβαίως δεν συμπεριφέρονται πάντα όπως θέλουν τα μοντέλα. Äh, Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις εντελεχείς ε, απαντήσεις. Σίγουρα είναι πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά που είπατε ότι ένα μοντέλο εν γέννη δεν μπορεί ποτέ να είναι 100% ακριβές. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει, και εδώ δίνω δίκιο στους συναδέλφους, μέχρι στιγμής πάντα εμφανιζόταν σαν να ήταν κατά κάποιο τρόπο το σίγουρο, κάτι το οποίο ήταν πολύ σαφές ότι από αυτό το μοντέλο βγαίνουν σαφή αποτελέσματα και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια διαφοροποιημένη αντιμετώπιση, να δούμε τι λένε άλλα μοντέλα και αυτό που λένε οι συνάδελφοι προφανώς έχει συνέπειες για τις ε, ε, συνέπειες, το αν είναι οι συνέπειες που πρέπει να εξαχθούν από αυτό το μοντέλο. Οι συνάδελφοι βέβαια είναι θεμητό να έχουν κάποιες εμφιβολίες αν είναι μονόδρομος τα αποτελέσματα αυτού του, του μοντέλου. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν κάποιο από την Επιτροπή που ξέρει καλά το μοντέλο να έρθει και να μα εξηγήσει περισσότερο. Πάντω όλα αυτά που είπατε ήταν πολύ ενδιαφέροντα θα σκεφτούμε για το αν θέλουμε να δώσουμε συνέχεια. Τώρα δεν υπάρχει ένα κάποιο άλλο ερώτημα. Μήπως μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο προς το παρόν. Έχουμε εμβαθύνει στο θέμα αυτό. Έχουμε θέσει ερωτήματα, έχουμε πάρει απαντήσεις και γι' αυτό νομίζω ότι αρκετό χρόνο χρησιμοποίησαμε. Μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο σας ευχαριστώ. wir dann indem wir jetzt... Προχωρούμε λοιπόν ερχόμαστε στην συζήτηση με τους δύο εμπειρογνώμονές μας για ένα συγκεκριμένο και επακριβές ερώτημα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι και οι δύο παρόντες εντάξει και έχουν παρακολουθήσει την ε, συζήτηση μέχρι στιγμής. Jetzt müssen Sie ihn anders oh,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 έχουμε καθαρίσει εδώ πέρα τα έδρανα. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στη συζήτηση με τον κύριο Άιχάμερ και τον δόκτορα Βάιμαν, τους δύο δόκτορες, τον καθηγητή μάλλον Βάιχμα και τον δόκτορα Άιχάμερ. Τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους και τη διαθέσιμό τους να είναι παρόντες για αυτή τη συζήτηση. Χαιρόμαστε που ήρθατε παρά το σύντομο χρονικό διάστημα που υπήρξε μετά την πρόσκλησή σας και πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αφορά την έννοια της έντασης ενέργειας δεν χρειάζεται να σας ε, παρουσιάσω. Στους φακέλους υπάρχουν τα, τα βασικά σας βιογραφικά στοιχεία. <laughs> Προσοχή για τη στάζει από παντού. Ωραία. Να ξεκινήσουμε τώρα τα πρότεινα. Κύριε Άιχ Χάμερ. Είχαμε συμφωνήσει λοιπόν να υπάρξει μια σύντομη παρουσίαση και μετά να προχωρήσουμε στην ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων. Καλό απόγευμα κυρίε και κύριοι. Wolfgang Eichhammer λέγομαι. Είμαι ερευνητή στο Ινστιτούτο Φράνχοφερ στη Γερμανία και έχω εμπλακεί σε διάφορα επίπεδα, σε διάφορα στάδια στην οδηγία ενεργειακής απόδοσης από το 2006 και σε κάποιο βαθμό και στην αξιολόγηση για την προτινόμενη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Αυτό το οποίο μου ζητήθηκε είναι να απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα και να κάνω κάποιες δηλώσεις και όλα αυτά τα συνοψίζω εδώ. Ένα πρώτο ερώτημα είναι πώς πρέπει να καθορίσουμε τους στόχους ενεργειακής απόδοσης υπάρχει μια συζήτηση σε σχέση με απόλυτους στόχους αποδοτικότητας και άλλοι υποστηρίζουν πρέπει να ακολουθήσουμε σχετικούς στόχους. Δεν θέλω να αντιμετωπίσω το ερώτημα του αν οι στόχοι οι οποίοι προτείνονται στην οδηγία περιορίζουν την οικονομική ανάπτυξη, αν η φιλοδοξία του θα πρέπει να αλλάξει μέσα στα πλαίσια οικονομικής κρίσης ή ισχυρής μεγέθυνσης, πόσο πολύπλοκη είναι η ισχυρης μεγεθυνση ποσο παρακολούθησης, πώς θα μπορέσει να γίνει κατανομή προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών και ποια είναι τα κύρια μηνύματα την σηματοδότηση από την ε, διατύπωση μάλλον του στόχου. Πρώτο ερώτημα. Πώς καθορίζουμε τους στόχους, πώς ορίζουμε τους στόχους εξοικονόμηση ενέργειας. Ένας τρόπος είναι να συγκρίνουμε με ένα συγκεκριμένο έτος. Παραδείγματος χάρη το 2007. Και ο στόχος θα μπορούσε να διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε σε σχέση με το 2007 η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας να μειωθεί κατά 20% μέχρι το 2020. Επομένως, μια μείωση κάτω το, από το σημερινό επίπεδο. Και αυτό είναι παράλληλο, είναι παρόμοιο με τους στόχους του Κιώτο για τα αέρια θερμοκηπίου. Αντίθετα τώρα υπάρχει μια πρόταση από την Κομισιόν στην προτινόμενη οδηγία. Αυτό δεν είναι σε σχέση, ο στόχος αυτός δεν είναι σε σχέση με ένα συγκεκριμένο έτος, αλλά λαμβάνει υπόψη και την οικονομική ανάπτυξη από σήμερα μέχρι το 2020. και είναι μια ε, μείωση σε σχέση με το προσδοκόμενο επίπεδο κατανάλωσης το 2020. Επομένως είναι μεγαλύτερη η μείωση από αυτήν που αναφέρεται στο γράφημα αριστερά. Αυτό αναφέρεται λοιπόν σαν πρόταση από την Κομισιόν. Και υπάρχει και μια άλλη αντιμετώπιση, ένα στόχος για την ένταση εργασίας, έχουμε μια συγκεκριμένη ένταση εργασίας σήμερα, η οποία μειώνεται με το χρόνο, με αυτόνομη δυναμική, αλλά λόγω και των μέτρων πολιτικής τα οποία υλοποιούνται. Και εκεί μπορεί να διατυπωθεί ένα στόχος σε σχέση με το επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να μειωθεί η ένταση ενέργειας. Το κύριο πλεονέκτημα ενός στόχου έντασης ενέργειας είναι ότι καταρχήν είναι ανεξάρτητος αυτός ο στόχος από το επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας και αυτό είναι φυσικά και το πρόβλημά του γιατί η ανάπτυξη της οικονομικής ανάπτυξης μπορεί να αναστρέψει τα κέρδη από την αύξηση της, από τη μείωση της έντασης ενέργειας. Ο στόχος που προτείνεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζει την οικονομική ανάπτυξη, εγώ θα έδινα την απάντηση, απάντηση όχι. Και εδώ και στην επόμενη διαφάνεια είναι οι απαντήσεις. Ο πρώτος στόχος είναι ότι ο στόχος βασίζεται στα αποτελέσματα του Primes για το 2007 και που είναι η βάση για τη διατύπωση των στόχων ήταν μια, ένα σημείο αναφοράς πριν από την οικονομική κρίση και βασίζεται σε ένα σενάριο 2,4% οικονομικής ανάπτυξης κατά μέσο όρο μεταξύ 2005 και 2020. Τώρα είμαστε παρασάγκα μακριά από το 2,4% ως ε, μέσο όρο. Αν δείτε λοιπόν τις προβλέψεις που είναι διαθέσιμες μέχρι το 2013, μπορείτε να Φανταστείτε ότι χρειάζεται μία θαυματουργή μεγέθυνση 4% στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φτάσουμε το σημείο στο οποίο ο στόχος του 20% θα περιορίσει την οικονομική μεγέθυνση. Μόνο δηλαδή αν ξεπεράσουμε μία μεγέθυνση 4% το χρόνο θα είναι περιοριστική η στόχη της ενεργειακής ε, έντασης σε σχέση με αυτό που είχε επιτευχθεί το 2007. Αυτό είναι σαφές στην ε, σύγκριση αυτή φαίνεται ο ιστορικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ με την μπλε γραμμή και η κόκκινη γραμμή δείχνει το 4% που θα είναι απαραίτητο για, από το 2012 στο 2020 για να φτάσουμε τα όρια της ανάπτυξης και βλέπετε ότι τα τελευταία 20 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πετύχει σχεδόν ποτέ ένα τόσο φιλόδοξο στόχο 4% μεγέθυνσης. Το επόμενο ερώτημα. Η φιλοδοξία του στόχου αλλάζει μέσα στα πλαίσια μιας οικονομικής κρίσης, μιας ταχείας οικονομικής μεγέθυνσης. Το κύριο μήνυμα, μήνυμά μας είναι ότι ένας στόχος κατανάλωσης, απόλυτος στόχος δηλαδή που να περιλαμβάνει και τη μεγέθυνση, είναι πολύ πιο εύκολο να εκπληρωθεί σε καιρούς οικονομικής κρίσης και λιγότερο εύκολο να επιτευχθεί σε καιρούς μεγάλης οικονομικής μεγέθυνσης. Ενώ ένας στόχος ένταση είναι πιο δύσκολος να επιτευχθεί όταν είναι αργή η οικονομική ανάπτυξη και ευκολότερο να επιτευχθεί όταν είναι υψηλή η οικονομική ανάπτυξη. Πηγαίνουν λοιπόν αντίθετα στα αποτελέσματά τους αυτές οι δύο στοχοθεσίες. Το να μεταφέρει κανείς τον στόχο της κατανάλωσης σε ένα στόχο έντασης είναι κάτι που θα καταστήσει πιο δύσκολη την κατάσταση σε σχέση με τις συνθήκες χαμηλότερης οικονομικής ανάπτυξης σήμερα. Εδώ βλέπετε την αύξηση του ΑΕΠ, όταν είναι χαμηλή η αύξηση αυτή, Βλέπετε ότι όταν ε, η αύξηση του ΑΕΠ είναι υψηλή, τότε η ενέργεια αυξάνεται πιο γρήγορα και όταν επιβραδύνεται η αύξηση του ΑΕΠ, τότε και η ενέργεια μειώνεται λιγότερο γρήγορα και πολλές φορές είτε αυξάνεται είτε μένει στάσιμη. Αυτό ίσως να σημαίνει κάτι ότι η αποδοτικότητα της ενέργειας είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πετύχουμε με χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Από την άλλη, όταν εξοικονομούμε ενέργεια, όπως βλέπουμε στη μελέτη, αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα όταν σοβεί μια οικονομική κρίση. Το επόμενο θέμα για έναν στόχο κατανάλωσης που να συμπεριλαμβάνει την οικονομική ανάπτυξη είναι η περιπλοκότητα της διαδικασίας εποπτείας, ελέγχου αν θέλετε. Αυτό έχει φανεί από τις συζητήσεις που έγιναν από το 2006 για την τότε οδηγία, όταν δημιουργήθηκε μια νέα διαδικασία απαρακολούθησης και συνέχειας, αν θέλετε, της κατάστασης και κατά κάποιο τρόπο λειτουργήσε ε, παραπλανητικά σε σχέση με τους βασικούς στόχους τους οποίους είχαμε. Ο στόχος της κατανάλωσης είναι κάτι το εύκολο καταρχάς, διότι χρειάζεται απλά ένας απολογισμός σε σχέση με τη χρήση της ενέργειας. Απ' την άλλη, αν έχει κανείς την ένταση, πρέπει να δει και τα επιπλέον στοιχεία δραστηριότητας, και σε σχέση με το ΑΕΠ και αυτό είναι κάτι το οποίο κυμαίνεται πολύ περισσότερο από ότι η κατανάλωση της ενέργειας και καθιστά όλα τα στατιστικά στοιχεία πολύ περισσότερο αβέβαια. Το θέμα είναι πώς μπορεί να υπάρξει η κατανομή της προσπάθειας ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η σήμερα κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ήδη λαμβάνουν υπόψη την κατανομή της προσπάθειας μέσω της στρατηγικής 2020. Σαν παράδειγμα, κάποιες ε, χώρες ε, ε, της Ανατολικής Ευρώπης, Ανατολικής Ευρώπης έχουν θα έλεγα μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης σε κάποιους βασικούς τομείς, αλλά όχι σε άλλους τομείς. Πάντως βλέπουμε ότι πολλές ανατολικές χώρες είναι υψηλότερα από ό,τι χώρες όπως η Γερμανία. Η συζήτηση σε σχέση λοιπόν με την κατανομή του βάρους ε, και της προσπάθειας έχει ήδη προχωρήσει. Απαιτούνται όμως νέα σετ δεδομένων, απαιτούνται νέες συζητήσεις για την κατανομή της προσπάθειας κάτι το οποίο δυστυχώς θα προκαλέσει ακόμα περισσότερες καθυστερήσεις στη διαδικασία ορισμού στόχων για τα μεμονωμένα κράτη-μέλη και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε το 2014. Έρχομαι στην τελευταία διαφάνεια και στο τελευταίο μήνυμα, αν θέλετε, το οποίο θα ήθελα να σας μεταφέρω για τη διατύπωση, τη σωστή μορφοποίηση του στόχου και για την κατανάλωση και για την ένταση. Καταρχάς ο στόχος κατανάλωσης βοηθάει στη συνειδητοποίηση της αγοράς νέγκαβατ και βάζει αν θέλετε κάποια επιπλέον κίνητρα προς τις κυβερνήσεις για να αναπτύξουν τις υπηρεσίες ενέργειας στην ουσία υπάρχουν και κάποιες άλλες πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές σαν παράδειγμα που συμβαδίζουν. Και εφόσον έχουμε σαν τελικό στόχο τη μείωση κατά 80% πρέπει η προσπάθειά μας να είναι πάρα πολύ συστηματική και συνειδητή. Και στις υποδομές και στις γραμμές μεταφοράς, τα δίκτυα μεταφοράς. Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν αυτές τις υποδομές και αν αυτές οι υποδομές μπορεί να αποφευθούν και το κόστος φυσικά το οποίο συνεπάγονται, τότε θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε οι στόχοι αυτοί να μπουν πολύ πιο εύκολα στις νοοτροπίες και στους στόχους. Το τρίτο μήνυμα, στα πλαίσια της μορφοποίησης του στόχου θα έλεγα, είναι ότι ο στόχος της κατανάλωσης λαμβάνει υπόψη και κάποιες, κάποιες αναπηδήσεις οι οποίες δεν καλύπτονται στην κατανάλωση, που δεν καλύπτονται από τους στόχους έντασης. Όσο ο κόσμος εξοικονομεί ενέργεια και εξοικονομούνται χρήματα, τότε χρησιμοποιούνται χρήματα για ενέργεια σε άλλους τομείς. Αυτό είναι ένα παράπλευρο φαινόμενο. Και τέλος, η μείωση της ενέργειας σε απόλυτους όρους ε, θέτει την ανάγκη αν θέλετε ενός απόλυτου στόχου και δημιουργεί δυνατότητες και για αύξηση του ΑΕΠ και για αύξηση των θέσεων απασχόλησης και για αύξηση σε επενδύσεις ε, μειώνοντας το κόστος της ενέργειας σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου. Ευχαριστώ. Herr Professor Weimann, Sie sind am Zuge καθηγητά. Ja, και κύριοι, πριν ξεκινήσω την παρουσίασή μου, επιτρέψατε μου δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση αφορά ε, το τι είμαι εγώ. Είμαι οικονομολόγος, οι οικονομολόγοι βέβαια έχουν άσχημη φήμη όταν ασχολούνται με ε, ζητήματα περιβάλλοντος. Γι' αυτό, καλό θα ήταν να σα πω ποιο είναι το ενδιαφέρον μου. Είμαι οικονομολόγος του περιβάλλοντος και εγώ θα ήθελα να συνεισφέρω να χρησιμοποιούμε καλύτερα τους ε, λίγους πόρους που έχουμε για την κλιματική αλλαγή για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην τεράστια αυτή πρόκληση. Οπότε θέλω να βρω τα καλύτερα μέσα ε, που μπορούμε να έχουμε για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, γιατί θεωρώ πως μόνο αν γίνει αυτό έχουμε μία πιθανότητα. Τη δεύτερη παρατήρηση, η δεύτερη παρατήρηση. Με προσκάλεσαν τελευταία στιγμή και δεν ήξερα τι να περιμένω. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω κάποιες γενικές έτσι, σκέψεις πιο γενικές από αυτές του συναδέλφου που ίσως να σας φαίνονται και κάπως ασήμαντες αλλά χρειάζεται να κάνω αυτή την εισαγωγή για να καταλήξω στην πρότασή μου. Για να δούμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ απολύτων και σχετικών στόχων. Αυτά ως παρατηρήσεις. Αυτές ήταν. Δηλαδή, παρατηρήσουμε παρατηρήσει μου, οπότε παρακαλώ να ξεκινήσει από τώρα μετράει ο χρόνος μου. Λοιπόν, να θα παρουσιάσουμε κάποιες απλές σκέψεις για τη χρήση της ενέργειας. Χρησιμοποιούμε ενέργεια γιατί θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, όχι να σπαταλάμε ενέργεια. Στέλνουμε τα σπίτια μας, το νερό και τα λοιπά. Οπότε αφενός έχουμε την ε, ίδια την ενέργεια ως πόρο και από το τι θα επιτύχουμε με αυτήν. Οπότε όταν μιλάμε για εξοικονόμηση πρέπει να λάβουμε υπόψη τις δύο αυτές πτυχές. Οπότε αν μιλάμε για εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να γνωρίζουμε πως έχουμε κάποια οικονομία αλλά συμβαίνει και κάτι άλλο. Δηλαδή το κόστος το οποίο δημιουργείται από αυτή την εξοικονόμηση και πάει χέρι με χέρι μαζί της. Το κόστος αυτό προκύπτει είτε από το ότι δεν επιτυγχάνουμε τους στόχους όσο θα θέλαμε ή όσο τους επιτυγχάναμε πριν, γιατί υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, με το κόστος ευκαιρίας δηλαδή, ή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλους πόρους για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με λιγότερη ενέργεια. Να χρησιμοποιήσουμε πόρους δηλαδή για να αντισταθμίσουμε την ε, απώλεια της ενέργειας. Ανεξάρτητος του τι κάνουμε λοιπόν, πρέπει πάντα να υπολογίζουμε την αντιστάθμιση αυτή αφενός, δηλαδή την εξοικονόμηση ενέργειας και το κόστος που προκύπτει από την άλλη. Φαίνεται βεβαίως κάτι ασήμαντο. Και λέτε γιατί το λέει αυτός. Σκεφτείτε το εξή και ίσως δεν σας φαίνεται τόσο ασήμαντο. Πρώτον το ερώτημα. Δεδομένου αυτού είναι καλή στρατηγική να λέμε όπως λέει η οδηγία δηλαδή εδώ πέρα για την οποία μιλάμε θα εξοικονομήσουμε 20% ενέργεια χωρίς να μιλήσουμε για το κόστος που θα δημιουργηθεί και χωρίς να ορίσουμε κάποια μέτρα για να φροντίσουμε να έχει ελάχιστο κόστος αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι ρητορικό βεβαίω το ερώτημα γιατί αν το κάνουμε αυτό δεν είναι καλή η στρατηγική γιατί διατρέχουμε τον κίνδυνο να γίνει μια εξοικονόμηση ενέργειας η οποία θα είναι παράλογη γιατί υπάρχουν εναλλακτικέ οι οποίες με λιγότερο κόστος θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. Αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει πω θα μπορούσαμε να ε, έχουμε λιγότερη εξοικονόμηση ενέργειας. Δηλαδή η εξοικονόμηση την οποία θα κάνουμε χωρίς να λάβουμε υπόψη το κόστος θα είναι οπωσδήποτε μικρότερη από αυτή την οποία θα μπορούσαμε δυνητικά να επιτύχουμε. Το δεύτερο ερώτημα είναι χρειάζομαστε το κράτος όταν μιλάμε για το να ζυγίσουμε το κόστος ε, και την εξοικονόμηση ενέργειας. Όχι απαραίτητα. Θα μπορούσε κανείς πρώτα απ' όλα να πει πως οι αγοράες ενέργειας κάνουν ήδη καλά τη δουλειά τους. Υπάρχουν τιμές ενέργειας και οι καταναλωτές και οι επιχειρηματίες στην Ευρώπη έχουν κάθε λόγο να ζυγίσουν πολύ προσεκτικά το εάν είναι δυνατόν να εξοικονομήσουν ενέργεια με χαμηλό κόστος και αν προκύπτει ένα εκτιμά. Και μπορούμε να το προχωρήσουμε ακόμη περαιτέρω και να πούμε εντάξει εν μέρη στις τιμές στις οποίες έχουμε στις αγορές ενέργειας υπάρχουν ήδη τόσο πολλοί φόροι ε, και υπάρχει ήδη ενσωματωμένο το κόστος του διοξιδίου του άνθρακα ώστε μπορούμε να πούμε πως ε, έχουμε ενσωματώσει το εξωτερικό κόστος. Οπότε δεν είναι εκ των προτέρων σαφές το γιατί χρειάζεται κρατική ρύθμιση για να αυξηθεί η ενεργειακή αποτελεσματικότητα ή να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Η μόνη λογική εξήγηση για κρατική παρέμβαση είναι πως υποθέτουμε πως τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις συστηματικά αγνοούν σημαντικές στοιχές της χρήσης ενέργειας ή τουλάχιστον δεν λαμβάνουν υπόψη είναι όπως εμείς θα θέλαμε. Το ερώτημα είναι ποιες πτυχές θα μπορούσαν να είναι αυτές. Και εδώ πέρα ε, απαντάει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις προκλήσεις που θέλει να απαντήσει. Πρώτα απ' όλα η διασφάλιση της προμήθειας ενέργειας, με το οποίο εννοούμε αφενός πρόσβαση σε πηγές ενέργειας και βεβαίως από την άλλη εννοούμε και την ε, π.χ. να είναι σίγουρα και ασφαλή τα ηλεκτρικά δίκτυα. Δεύτερη πρόκληση είναι η αηφορία που μιλάμε εκεί για την προστασία πρώτα απ' όλα των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τρίτον, βεβαίως, είναι η προστασία του κλίματος, κάτι το οποίο είναι ταυτόσιμο με τη μείωση των εκπομπών. Και τέταρτο, που ορίζει η Κομισιόν, είναι η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και άρα αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι χαμηλές τιμές σε σχέση με τη διεθνή σύγκριση. Εάν δούμε αυτούς τους στόχους, θέλω άρα να ξαναθέσω το ερώτημα. Είναι λογική συμπεριφορά και απάντηση σε αυτούς τους τέσσερις στόχους και προκλήσεις να πούμε και να απαιτήσουμε ε, να μειώσουμε την ε, κατανάλωση ενέργειας κατά 20% ε, τις 100 χωρίς να λάβουν υπόψη το κόστος που θα προκύψει ε, από αυτές. Δεν είναι, δεν είναι λογικό. Και για να το δούμε θα ήθελα να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Το οποίο συνοψίζει δύο προκλήσεις, η μία είναι η αεφορία και η άλλη είναι η προστασία του κλίματος. Γιατί αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κλίμα, αυτό γίνεται με την ε, μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του ε, άνθρακα, πλην βεβαίω τη δέσμευση και αποδίκευση άνθρακα. Άρα αυτό σημαίνει μείωση των ορικτών καυσίμων. Άρα μιλάμε ειδικά για τα ορικτά ε, καύσιμα. Οπότε αυτοί οι δύο στόχοι είναι μαζί. Αν θέλετε είναι ένας και ο ίδιος Ας δούμε λοιπόν αυτό το θεμελιώδες ε, θέμα. Θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε τις εκπομπές. Το πρόβλημα είναι πως γνωρίζουμε πως αυτό κοστίζει. Είναι γενικώ γνωστό. Γνωρίζουμε επίσης πως οι πόροι τους οποίους έχουμε για να το κάνουμε αυτό είναι Περιορισμένοι. Μπορούμε λοιπόν να συζητήσουμε πόσους πόρους θα χρησιμοποιήσουμε γι' αυτό και η απάντηση ε, σε κάθε χώρα είναι διαφορετική, αλλά ανεξαρτήτως του πώς γίνεται αυτή η συζήτηση, στο τέλος θα προκύψει πως ε, έχουμε περιορισμένους πόρους. Και αυτό το οποίο χρειαζόμαστε άρα είναι λίγη λογική. Δηλαδή, εάν συνοψίσουμε αυτά τα τρία πράγματα προκύπτει μοιραία πως μόνο μία αποτελεσματική ως πρώτο κόστος πολιτική μείωση του οξυδίου του άνθρακα είναι λογική. Αυτό σημαίνει πως ε, αποτελεσματικότητα ως πρώτο κόστος σημαίνει μεγιστοποίηση των τόνων διοξιδίου του άνθρακα που μειώνονται ανά εκατομμύριο ευρώ επένδυση ή αλλιώ ελαχιστοποίηση του κόστους ε, του οριακού, του ενός επιπλέον τόνου διοξιδίου του άνθρακα. Αν παραμελούμε αυτόν τον απλό κανόνα, αυτό σημαίνει μοιραία πως σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα από ό,τι θα μπορούσαμε ιδεωδώς με τους πόρους μας. τι σημαίνει αυτό, σημαίνει κάτι πολύ απλό. Αν αυξήσουμε την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, τότε είναι μία αναγκαία συνθήκη αυτό για να έχουμε μία λογική κλιματική πολιτική. Αλλά δεν είναι επαρκής. Είναι αναγκαία και ικανή μόνο εάν από τις πολλές δυνατότητες που υπάρχουν επιλέξουμε εκείνες οι οποίες κοστίζουν λιγότερο. Μόνο έτσι έχουμε μια λογική πολιτική κλίματος. Φανταστείτε να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα με τρόπο ο οποίος δεν θα είναι ιδεώδης από πλευράς κόστους. Ε, αυτό το οποίο θα δούμε είναι πως για την ίδια ποσότητα μείωσης με ε, αποτελεσματικό τρόπο θα είχαμε ε, με τα ίδια χρήματα επιτύχει πολύ μεγαλύτερη μείωση. Άρα αν παραμελούμε το κόστος αυτομάτως οδηγούμαστε στο ότι δεν επιτυχάνουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Πώς θα επιτύχουμε λοιπόν την ε, πολιτική αυτή με το ε, μικρότερο κόστος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πως έχει το τέλειο μέσο για αυτή τη δουλειά, δηλαδή το εμπόριο εκπομπών, το οποίο είναι ιδανικό για να επιτύχουμε όλους τους στόχους της κλιματικής πολιτικής. Γιατί? Συνδέει τα εξής και έχει τις εξής ιδιότητες. Με το πλαφόν ορίζουμε ακριβώς ποιες θα είναι οι κομπές που θέμα. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε για ολόκληρη την οικονομία. Αυτό σημαίνει πω ο περιβαλλοντικό στόχο που έχουμε μπορεί να οριστεί πολύ επακριβώς. Και αυτό μπορεί να γίνει για οποιονδήποτε άρα στόχο που θέλουμε. Δεν υπάρχει κάποιο περιορισμό. Το εμπόριο το οποίο ξεκινάει έτσι και η αγορά που υπάρχει χάρη σε αυτό μας εγγυάται πως οι μειώσει που γίνονται είναι πράγματι αποτελεσματικές ως προς το κόστος. Δεν έχω τον χρόνο τώρα να σας εξηγήσω το γιατί. Επιπλέον η αγορά αυτή έχει ένα άλλο πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, δηλαδή δημιουργεί κίνητρα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αποφυγής της εκπομπής. Οπότε έχουμε ένα μέσο το οποίο δημιουργεί κίνητρα υπό την έννοια πως ο κάθε δρόν έχει κίνητρο να αναπτύξει την τεχνολογία που χρειαζόμαστε όλοι. τεχνολογία δηλαδή που μειώνει τις εκπομπές. Και επιπλέον δεν απαιτείται άρα περαιτέρω παρέμβαση. Αντιθέτως, περαιτέρω παρέμβαση είναι αντιπαραγωγικές. Να το αιτιολογήσω και από τις δύο πλευρές. Από την πλευρά της προσφοράς έχουμε τις γνωστές τιμές για την προώθηση ε, της ανανεώσιμης ενέργειας. Αυτό δεν οδηγεί σε περαιτέρω μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, γιατί οποιαδήποτε μείωση μετά οδηγεί σε πώληση των ε, δικαιωμάτων εκπομπής. Εάν κάποιος άρα παράγει, ε, εκπέμπει λιγότερο. η ποσότητα εκπομπής αυτή, άρα γίνεται μόνο μέσω, ορισμό του πλαφών, μέσω του ορισμού του πλαφών, κυρίες και κύριοι. Το κόστος το οποίο προκύπτει τώρα, αν, αντικαταστη... αν μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακος με ηλιακή και ολική ενέργεια, το κόστος το οποίο προκύπτει είναι τεράστιο. Για ένα τόνο διοξείδιο του άνθρακος με ολική ενέργεια τον ε, αντικαταστήσουμε. Χρειάζεται 100 με 150 ευρώ τον τόνο και για την ηλιακή ενέργεια 500 με 1000 ευρώ. Επομένως, βλέπετε ότι αυτό είναι πολύ περισσότερο από το οριακό κόστος στην εμπορία εκπομπών με 15 με 20 τόνους, 20 ευρώ το τόνο. Η έκθεση Μπέργκερ και Ρόσενταλ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κόστος της μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος αυξάνεται λόγω της προώθησης των ανανεωσίμων ενεργειών. Βλέπετε εδώ λοιπόν το ποσοστό της χρήσης πρασίνων ενεργειών και το πρόσθετο κόστος το οποίο θα προκληθεί μέσα στο πλαίσιο αυτό το οποίο, στο οποίο έχει δεσμευτεί να, κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει λοιπόν ποιο είναι το κόστος συμμόρφωσης το οποίο περίπου διπλασιάζεται. Στην Γερμανία έχουμε ήδη τέσσερις φορές αύξηση του κόστους αν έχουμε μία μείωση κατά 18%. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σωστό η σωστή σχέση κόστους ωφέλειας. Επίσης με την ναι. Οι τιμέ λοιπόν για το διοξείδιο του άνθρακος αντιδρά λόγω της ε, πράσινη ενέργειας. Αυτό είναι κακό. Εμείς θέλουμε να είναι ψηλό το κόστος των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Βλέπετε λοιπόν ότι εάν είναι φτηνή η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος δεν λειτουργούν τα κίνητρα. Ουσιαστικά καταστρέφεται η παροχή κινήτρων με την ε, διαδικασία αυτή. Οπότε, εάν υπάρξει αύξηση της ε, πράσινης ενέργειας, θα μειώσει ακόμα περισσότερο την τιμή των πιστοποιητικών εκπομπής ενέργειας. Βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχει και μία επίπτωση στον κύριο φορέα ενέργειας στην Γερμανία. Βλέπετε ότι υπάρχει αύξηση της χρήσης λιγνίτη στην Γερμανία. Είναι όμως ο φορέας ενέργειας ο οποίος έχει το μεγαλύτερο επίπεδο εκπομπής διοξιδίου του άνθρακος και λόγω των χαμηλών τιμών διοξιδίου του άνθρακος αυξάνεται η χρήση λιγνίτη. Και το ίδιο ισχύει για την πλευρά της ζήτησης της αγοράς. Όταν δείτε τους κανονισμούς για την ε, αποδοτικότητα της ενέργειας από την πλευρά της ζήτησης, βλέπετε ότι τέτοια πράγματα γίνονται. Η μείωση διοξιδίου του άνθρακος που προέρχεται από αυτούς τους κανισμούς οδηγεί σε μια ανακατανομή και όχι σε μια μείωση των δικαιωμάτων εκπομπής. Το κόστος λοιπόν συμμόρφωσης αυξάνεται και πάλι. Τι μπορώ να καταλήξω, τι μπορώ να καταλήξω. Οποιαδήποτε πολιτική η οποία προσπαθεί να μειώσει τις εκπομπές κάτω από το όριο το οποίο έχει καθοριστεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καταρχήν ε, περιττή, δεύτερον αυξάνει το κόστος και τρίτον μειώνει την συνολική αποδοτικότητα ενέργειας. Είναι μικρότερη λοιπόν η αποδοτικότητα της ενέργειας που θα μπορούσε να επιτευχθεί. Και έρχομαι τώρα στο κύριο ερώτημά σας. κατά πόσο η οδηγία για την ενεργειακή εξοικονόμηση θα πρέπει να θέσει απόλυτους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας ή αν θα πρέπει να αναφέρει στόχους σχετικής αποδοτικότητας, δηλαδή τόνους κατά εκατομμύριο ευρώ ΑΕΠ. Ένα άλλο σημείο το οποίο έχει σημασία στη συζήτηση, από ό,τι είδα, είναι και το ερώτημα τι είδους ρυθμίσεις, τι μορφή ρυθμίσεις είναι καλύτερη για την οικονομική ανάπτυξη. Και αυτό το ανέφερε και ο κ. Χάμερ. Αν το δούμε λοιπόν σε ένα πίνακα και δούμε ποια εργαλεία είναι τα πιο κατάλληλα για κάθε κατάσταση ή απόλυτος στόχος ή στόχος ε, αποδοτικότητας σχετικό σε περίοδο οικονομικής ανάπτυξης ή σε περίοδο ύφεσης, σε περίπτωση ε, οικονομικής ανάπτυξης θα υπάρξει μεγαλύτερη ε, ανάπτυξη από το στόχο της ανάπτυξης, ενώ σε μία ύφεση είναι πιο εύκολο να βγει κανείς από την ύφεση όταν έχει ένα απόλυτο στόχο παρά όταν έχει ένα σχετικό στόχο. Είδατε και από τα στοιχεία του κυρίου Άιχ Χάμερ ότι σε μια περίοδο ύφεση η μειώνεται η αποδοτικότητα ενέργειας. Άμα πέσουμε λοιπόν σε μία φάση ύφεση, αν έχουμε ένα σχετικό στόχο, θα είναι μεγαλύτερος, μεγαλύτερο το κόστος επίτευξης της αποδοτικότητας. Αυτό δεν βοηθάει λοιπόν. Γι' αυτό είναι καλύτερα να έχει κανείς ένα απόλυτο στόχο παρά ένα σχετικό στόχο. Βλέπετε λοιπόν ότι Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν δεν είναι εύκολο να καταλήξει κανείς σε συμπεράσματα σαφή. Γι' αυτό κάνω μία πρόταση συμβαστή για ένα τρίτο δρόμο που λέει το εξής. Η συμβαστή λοιπόν αυτή λύση σημαίνει ο στόχος εξοικονόμησης κατά 20% θα πρέπει να μεταφραστεί σε αντίστοιχες μειώσεις εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Αυτό είναι εύκολο να το κάνουμε γιατί έχουμε ένα συγκεκριμένο μείγμα πρωτογενών φορέων ενεργείας. Βλέπουμε για να μειωθεί κατά 20% η κατανάλωση ενέργειας ποια θα είναι η μείωση του εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Μετά θα μειώσουμε το ανώτατο όριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα και έτσι με τον τρόπο αυτό οι συνέπειε είναι ότι μείωση κατά 20% στην ένταση ενέργειας που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη θα επιτευχθεί με αποκλειστικά, με τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, το οποίο είναι πολύ λογικό για την προστασία του κλίματος. Επιπλέον, λόγω της ε, διαδικασίας εκπομπής ε, εμπορίας εκπομπών θα υπάρξει μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε μη σπατάλη πόρων, θα γίνει με ένα αποτελεσματικό ως προς το κόστος τρόπο, δηλαδή θα μεγιστοποιήσουμε την αποδοτικότητα ενέργειας, θα την μεγιστοποιήσουμε μάλιστα. Και τελικά η διαδικασία αυτή της ελαχιστοποίησης του, κόστους θα είναι χρήσιμη και στην περίπτωση της περίοδου ανάπτυξης και στην περίοδο ύφεσης. Αυτή θα ήταν η πρότασή μου και ελπίζω ότι δεν σας ενοχλεί το ότι έκανα πολλές γενικές παρατηρήσεις και έδωσα αρκετά λίγο χρόνο σε αυτό το τελικό συμπέρασμα. Και σας ευχαριστώ για την προσοχή. Äh, Καταρχήν να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας και έρχομαι τώρα στη φάση των... της συζητήσεως ο κύριος Φόρντ. Κυρία Φόρντ έχει το λόγο. Πρώτη εσείς κυρία Φόρντ. No. No. Δεν θέλετε να μιλήσετε. Ο Τούρμες, κύριος Τούρμες. you two uh, contributions. Uh, I think... Ευχαριστώ και τους δύο μιλητές. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Έχουμε κάποιους στόχους στα πλαίσια αυτή της οδηγίας και το θέμα είναι αν οι στόχοι αυτοί είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Αν κατάλαβα καλά, ο στόχος ως έχει στην οδηγία είναι ένα σχετικό στόχος και όχι απόλυτος. Δεν ξέρω αν αυτό από μόνο του είναι μια απάντηση. Υπάρχει μια κάποια σύγχυση θα έλεγα στις συζητήσεις μας γιατί πολλοί πιστεύουν ότι ο στόχος της Επιτροπής είναι απόλυτος στόχος. ενώ στη συζήτηση φαίνεται ότι είναι ένας σχετικός στόχος γιατί αναφέρεται σε κάποια σενάρια και όχι γενικότερα σε σταθερούς αριθμούς. Από τις δύο ομιλίες βγαίνει το ότι αν θέλουμε να περάσουμε σε ένα στόχο έντασης της ενέργειας, αυτό σημαίνει ότι σε εποχές ύφεσης και μη αντίστοιχης απόδοσης της οικονομίας, ο στόχος θα είναι πάρα πολύ δύσκολα επιτεύξιμος. Θα, ενώ θα ήταν πολύ πιο εύκολος σε περίπτωση περίοδου με οικονομική ανάπτυξη. Κάποια λόμπι και κάποιες κυβερνήσεις πιστεύουν ότι θα πρέπει να βάλετε και κάποια άλλα χαρακτηριστικά στην πρότασή σας. Κάποιοι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά θα πιέσουν ακόμα περισσότερο την οικονομία από ότι αν εμέναμε στον βασικό στόχο της οδηγίας. Και τέλος για τον κύριο Βάιμαν. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αν πράγματι προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να μας εξηγήσετε γιατί είναι σημαντικό να υπάρξουν επιπλέον μετρήσεις και ανάλογα με τις μετρήσεις αυτές να υπάρξουν και οι ανώτατα, ενώτατα, ο καθορισμός των ανώτατων επιπέδων κατανάλωσης. Κύριος Βίλα Κουάδρας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόσφατα είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την οδηγία σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση και είχαμε κάνει τότε ήδη μια συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πιο πολύ σε φιλοσοφικό επίπεδο παρά σε οικονομικό επίπεδο για το αν θα ήταν καλύτερα να έχουμε σαν στόχο μια αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή αν θα έπρεπε να έχουμε σαν στόχο μια μείωση σε απόλυτους όρους της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Με μεγάλη προσοχή άκουσα αυτά που είπανε οι ομιλητές του απογέματος, ιδίως του κυρίου Άιχ Χάμερ, που εστιάστηκε στο τόσο ενδιαφέρον αυτό φιλοσοφικό σημείο και τα συμπεράσματα στα οποία φτάνω αφού έχω ακούσει τους δύο ομιλητές είναι τα εξής. Ελέγχθη ότι είναι πιο εύκολο να φτάσουμε σε απόλυτους όρους μείωσης της ε, ενεργικής κατανάλωσης όταν υπάρχει ύφεση. Ναι, ε, βέβαια. Και είναι πιο δύσκολο να το κάνουμε αυτό όχι, μάλλον, ότι είναι πιο εύκολο να το κάνουμε όταν υπάρχει ύφεση εννοώ και πιο εύκολο να το κάνουμε όταν πιο, πιο δύσκολο να το κάνουμε όταν έχει, υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να πετύχουμε ένα στόχο όταν αυταπατώμεθα. Έχουμε δηλαδή εκατομμύρια ανέργων που δεν καταναλώνουν αυτό που η οικονομία δεν παράγει, η βιομηχανία δεν παράγει και έτσι όπως είναι φυσικό ακόπως πετυχαίνουμε το στόχο της μείωση κατανάλωση πρωτογενού ενέργειας, όχι γιατί είμαστε πιο αποτελεσματικοί, αλλά γιατί είμαστε μπατήριδε, είμαστε πιο φτωχοί και δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε. Έτσι πιστεύω ότι το επιχείρημα ότι σε μία περίπτωση είναι πιο εύκολο δεν μου φαίνεται. Επειδή υπάρχει φτώχεια αυτό δεν μου φαίνεται ένα επιχείρημα το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο. Γι' αυτό εγώ ξαναλέω, επαναλαμβάνω αυτό το οποίο ότι χρειάζεται να ακούσουμε πιο πιστικά επιχειρήματα από αυτά που ακούσαμε σήμερα το απόγευμα και το λέω με κάθε ευγένεια ότι ο στόχος μας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα από τον υπάρχει ύφεση οικονομική ανάπτυξη να πετύχουμε μια μικρότερη κατανάλωση ενέργειας ενώ συγχρόνως θα έχουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Αυτή είναι η αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι καλό και σε στιγμές παχαίων αγελάδων και σε στιγμές ισχνών αγελάδων. Γιατί αυτό θα κάνει πιο ανταγωνιστική τη βιομηχανία μας και θα μπορέσουμε έτσι με τον τρόπο αυτό να προωθήσουμε τομείς που βασίζονται στην κατανάλωση ενέργειας και αυτό θα είναι και επίσης ένας τομέας της ενέργειας που θα δημιουργήσει νέες τεχνολογίες, θέσεις απασχόλησης, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις παγκόσμια αγορές Κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντική η παρουσίαση η οποία γίνεται. Κάποιες από τις ερωτήσεις που τέθησαν έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ο ορισμός της αποδοτικότητας της ενέργειας, η σχέση ανάμεσα στους στόχους, η σχετική στόχοι, οι απόλυτη στόχοι και ακόμα και οι παρατηρήσεις του κυρίου Τούρμες, ο οποίος εργάζεται για το θέμα αυτό, μας λέγει ότι κάποιοι από εμά που, κατα... που παρασκευάσαμε τις τροπολογίες δεν έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά το νόημα των στόχων, αν, είναι πρόκειται, αν πρόκειται για στόχους θα έλεγα σχετικούς ή απόλυτους. Γι' αυτό λοιπόν ένα αίτημα πρόεδρε. Θα προτιμούσα τέτοιες συναντήσεις να οργανώνονται κατά την αρχή της διαδικασίας γιατί στη συγκεκριμένη φάση αυτά τα που ακούμε βέβαια είναι πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα, αλλά θα προτιμούσα να τα άκουγα στην αρχή της διαδικασίας, στο ξεκίνημα. Ίσως λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε του χρόνου, όταν ξεκινήσουμε την αντίστοιχη διαδικασία και όχι τώρα που στην ουσία κλείνει η συζήτηση για τις τροπολογίες. Το σχόλιο μου ήταν λίγο τεχνικό αν θέλετε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σας το πω. Ακούγεται, δουλεύει, δουλεύει. Παράξενο μικρόφωνο είναι αυτό. Εγώ βρίσκω ενδιαφέρον που λέτε, αλλά εμείς πρέπει να οργανωθούμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Τα ερωτήματα βγαίνουν από την συζήτηση. Δεν υπάρχει ήδη από την αρχή το πλήρες φάσμα των ερωτημάτων. Έχετε ενδιαφέρον. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό στην αρχή ήταν πιο αποτελεσματικό, αλλά δεν υπήρχαν όλα τα ερωτήματα. Η κυρία λοιπόν Όλτς, την οποία ονόμασα λαθασμένα Φόρντ. Κυρία Χόλτ, συγγνώμη που, δεν, ε, που σας ονόμασα κυρία Φόρντ. Πάντα θα έχει ενδιαφέρον το να συζητάμε και διαφορετικές απόψεις και να ακούμε και τις απόψεις αυστηρά των οικονομολόγων. Θα ήθελα να μείνω λίγο σε αυτές τις απόψεις, σε κάποια σημεία τους, αλλά θα ήθελα να μείνω καταρχάς στις λεπτομέρειες στην, για την οδηγία αποδοτικότητας της ενέργειας. Όταν μιλάμε για το κόστος και το όφελος στα πλαίσια της οικονομίας, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσει κανείς ότι σε επίπεδο πρακτικής η μείωση της ενέργειας μπορεί να δημιουργήσει ωφέλη και όχι κόστος. Γιατί στην ουσία αυτό το οποίο πετυχαίνουμε, το πετυχαίνουμε και μέσω καινοτομιών, ξέρουμε, στα αυτοκίνητα, σε εξοπλισμού στο σπίτι και έτσι παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές με λιγότερη χρήση ενέργειας. Χάρη λοιπόν στην καινοτομία Υπάρχει μια ουσιαστική αποσύζευξη ανάμεσα στην χρήση της ενέργειας και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτά όλα θα δοκιμαστούν βέβαια στην αγορά και οι δυνατότητες τις οποίες έχουν οι μικτές μονάδες. Downing το θέμα είναι βέβαια να προσπαθήσουμε να δούμε αν στα πλαίσια της εμπορίας των εκπομπών οι αγορές μπορούν να αποδώσουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω τι θα πρέπει να κάνουμε, μήπως θα πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι πριν αποφασίσουν οι αγορές να αντιδράσουν. Για τις απόψεις του κύριου Άικαμερ. Ε, πείτε μου αν σας κατάλαβα καλά. Ανησυχείτε που αν, πως αν θέσουμε απλά και επιδιώξουμε το στόχο της έντασης, ο τρόπος για τις χώρες να τον πετύχουν είναι να διευρύνουν την παραγωγή τους. Και θα μπορούσαν να πετύχουν ένα τέτοιο στόχο έντασης της ενέργειας χωρίς να πάρουν κάποια μέτρα αλλαγής ουσιαστικά της πρακτικής τους. Και μας λέτε ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν χρησιμοποιώντας κάποιες καινοτομίες, κάποιες βελτιώσεις, αλλά όχι κάποιες αλλαγές ουσιαστικές. Τώρα σχετικά με την αύξηση του ΑΕΠ, δεν είναι υποχρεωτική η αύξηση της κατανάλωτης ενέργειας, και η μεθοδολογία παρόλα αυτά που ακολουθείτε δεν θα πρέπει να αλλάξει. Αν ακολουθήσουμε τη λογική αυτή, αυτές οι... αυτά τα παράσιτα ουσιαστικά τα οποία θα ακουστούν και χρησιμοποιήσατε τη λέξη παράσιτα για να μας πείτε ότι τα μέτρα αυτά θα επηρεαστούν πολύ από άλλου τύπου οικονομικές κυρίως δυνάμεις. Αυτά τα παράσιτα θα δημιουργήσουν αβεβαιότητα ως προς την επίτευξη των στόχων. Οπότε δεν καταλαβαίνω σε αυτή την περίπτωση πώς με τον στόχο έντασης της ενέργειας μπορούμε πράγματι να πετύχουμε ε, τον στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας, ούτε μάλλον να γνωρίζουμε αν θα τον πετύχουμε τον στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας, λόγω ακριβώς όλων αυτών των παρασίτων, θα έλεγα, στην αγορά. Ανησυχώ λοιπόν ε, για το τι θα συμβεί όταν ξεφύγουμε από, τις, από τους ρυθμούς της ύφασης, της ύφεσης. Η αλήθεια είναι ότι στη συγκεκριμένη φάση είναι εύκολο να μειώσει κανείς την ενέργεια, έτσι κι αλλιώς υπάρχει μικρότερη ζήτηση γιατί δεν υπάρχει ανάπτυξη οικονομική. Αλλά αν δεν επανεξετάσουμε θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε τις ενεργειακές υπηρεσίες, τότε δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά την ενέργεια και όταν βγούμε από την ύφεση και περάσουμε σε μια αναπτυξιακή περίοδο είναι σαφές ότι θα χρησιμοποιούμε τεράστιες ποσότητες ενέργειας μόνο και μόνο γιατί διαρθρωτικά δεν έχουμε κάνει αλλαγές. Είπατε επίσης και για τις λεγόμενες παραπλανητικές επενδύσεις. Ανησυχείτε για το κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει πάρα πολλές επενδύσεις που δεν θα πάνε τελικά προς τις ε, διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες θα πρέπει να γίνουν. Και αυτό γιατί δεν έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη για το πόση τελικά ενέργεια θα χρειαστούμε. Αυτό είναι κάτι που σας ανησυχεί αυτός ο στόχος που είναι λίγο θολός στον τομέα της έντοσης δεν μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα απώλειας επενδύσεων ή και ε, κακών στόχων, θα έλεγα λάθος στόχων στις επενδύσεις για την παροχή ενέργειας και, παροχή, και δημιουργία υποδομών για την παροχή ενέργειας τις οποίες δεν θα, δεν θα χρειαζόμαστε αλλά δεν θα γνωρίζουμε τον προτέρων αν χρειαζόμαστε ή όχι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τη συζήτηση αυτή τη θεμελιώδη θα δεν ήθελα εγώ να την έχουμε κάνει λίγο νωρίτερα. Όλοι όμως θεωρώ ότι θέλουμε να εξοικονομήσουμε πόρους και ενέργεια. Νομίζω πως χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία με το να ακολουθήσουμε χωρίς σκέψη την πρόταση της Κομισιόν. Σήμερα εγώ έμαθα πως υπάρχουν και μειονεκτήματα και με έναν απόλυτο και με έναν σχετικό στόχο. Έμαθα πως εάν επέκτηνε κανείς το σύστημα ε, εκπομπών ε, σε άλλους τομείς οικονομίας στα νοικοκυριά, παραδείγματο χάρη, θα γίνουν τα πιο απλά από τα 21 άρθρα που έχουμε τώρα. Όμω η οδηγία τώρα είναι αυτή που είναι. Πρέπει να εργαστούμε επ' αυτής. Και θα ήθελα να ρωτήσω του ειδικού. Μήπω μπορούμε να σκεφτούμε κάποιο συμβιβασμό, κύριε Βάιμαν. Ή κύριε καθηγητά, κύριε Άχημαν. Ένα σύνδεσμο μεταξύ απολύτου και σχετικού στόχου να το σχετίσουμε με, τους, με την συγκυρία που υπάρχει στην οικονομία και τον οικονομικό κύκλο ή μήπως να αφήσουμε ακόμη περισσότερο στα κρατη πώς θα επιτύχουν τους δεσμευτικούς στόχους που βεβαίως μπορούμε εμείς να ορίσουμε. Προέκυψε και η πρόταση αναφέρονται πιστοποιητικά και στην πρόταση μήπω μήπως το ETS, το σύστημα εμπορίας, να επεκταθεί σε εθνικό επίπεδο. Μήπως υπάρχει δυνατότητα να επιτύχουμε κάποιους συμβιβασμούς που θα καλύπτουν αυτές τις δυνατότητες που είδαμε σήμερα και να τις συνδέουν. Κυρία Τόγια. Ευχαριστώ. Κάποιες ερωτήσεις προς τον καθηγητή Αϊχάμερ. Δεν είμαι ειδικό στα θέματα της οικονομίας και δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς ίσως ορισμένα θέματα. Δύο πράγματα να ρωτήσω πάντως. Η σχέση ανάμεσα στους στόχους από τη μία και τις περιόδους χαμηλής ανάπτυξης όπως αυτή την οποία βιώνουμε. Είναι αλήθεια ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι και οι αναφορές της οδηγίας έχουν ισχύ θα έλεγα όταν αναπτύσσεται η οικονομία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι σε εποχές χαμηλής ανάπτυξης η επίτευξη συντεξιμένων στόχων δεν βοηθά την επανεκκίνηση του οικονομικού κύκλου. Γι' αυτό θα ήθελα να μου αποδείξετε το αντίθετο αν ισχύει. Είπατε επίσης ότι είναι πιο εύκολο να πετύχει κανείς τους στόχους της κατανάλωσης και όχι τόσο τους στόχους της έντασης σε εποχές χαμηλής ανάπτυξης, εξασθενημένης ανάπτυξης. Και για να περάσουμε από τον ένα στόχο στον άλλο απαιτείται πάρα πολύ χρόνος. Θα ήθελα λοιπόν να μας εξηγήσετε λίγο καλύτερα την ισορροπία ανάμεσα στις διαδικασίες επίτευξης των στόχων αυτών. Και επί τη βάση των πινάκων εδώ λέγεται ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα θεωρείται από την βιομηχανία ένα βάρος το οποίο θα πρέπει να άρει. Παρ' όλα αυτά η εξοικονόμηση η ενεργειακή μπορεί να ενισχύσει ακόμα και σε περίοδο κρίσης την ανάπτυξη και μάλιστα θα λέει κανείς ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης. Να μας πείτε λοιπόν ποια είναι τα δεδομένα τα οποία μπορεί να τεκμηριώσουν ένα τέτοιο ισχυρισμό και ίσως θα μπορούσαν τα συγκεκριμένα αυτά μέτρα να αναλυθούν καλύτερα ανά κράτος μέλος. Ίσως ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία να είναι καλύτερα προετοιμασμένα να εφαρμόσουν κάποιες μεθόδους οι οποίες να λειτουργήσουν παραδειγματικά και για τις υπόλοιπες. Υπόλοιπες που ίσως να σημειώνουν κάποια καθυστέρηση. Ο κύριος Ζαντό, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες, ιδίω η Φιώνα Χόλ, για την ποιότητα του μηνύματος που εμείς δίνουμε. Μπορεί κάντα, πάντα κανείς να ρωτάει για την ενεργειακή απόδοση. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι έχουμε προοδεύσει πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά καταναλώνουμε πάντα πολύ ενέργεια. Επομένως η ένταση εργασίας δεν σημαίνει και απόλυτη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό το έχουμε δει και στο παρελθόν. Μήπως μπορεί να είναι η λύση του μέλλοντος. <clears throat> Για μένα, σήμερα το μεγάλο πρόβλημα του βιομηχανικού μας συστήματος είναι η ποιότητα των μηνυμάτων που στέλνουν οι δημόσιες αρχές. Κατά την άποψή μου, στείλουμε το μήνυμα ότι που έχει να κάνει και με την αύξηση της οικονομικής, που έχει να κάνει μόνο με την αύξηση της ε, οικονομικής δραστηριότητας, δεν αποτελεί ένα σαφές μήνυμα για τις βιομηχανίες μας. Το μόνο σαφές μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε στις βιομηχανίες μας είναι ένας συγκεκριμένος στόχος δεσμευτικός για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Δεύτερο σημείο. Και εκεί έχει δίκιο ο Βιδαλ Βιδαλκουάδας. Είμαστε σε ύφεση. και η μείωση της κατανάλωσης είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας μείωσης εισοδημάτων. <clears throat> Μπορούμε να γυρίσουμε ανάποδα το επιχείρημα, αν στα επόμενα χρόνια, μας λέει ο Σάκη η Κομισιόν, θα έχουμε περιορισμένη μας λέει θα έχουμε περιορισμένη μεγέθυνση, αλλά α πούμε ότι ξαναγυρίζουμε σε μεγάλη οικονομική μεγέθυνση στι αναπτυγμένες χώρε. Η μεγέθυνση σημαίνει και αύξηση μηχανιστικά των τιμών ενέργειας. Και αυτό πάλι σημαίνει ότι γίνονται φτωχότεροι καταναλωτές. Και πάλι λοιπόν ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτό το διακύβευμα της αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων είναι να έχουμε ένα σαφές μήνυμα ότι πρέπει να μειωθεί σε απόλυτους όρους η κατανάλωση ενέργειας. Μόνο με τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας θα μπορέσουμε <clears throat> να μειώσουμε την, το λογαριασμό που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Για τον κύριο Χάμερ και τον κύριο Βάισμαν. Στην ανάλυση σας. Στην ε, ανάλυση σας έχετε και το συμπέρασμα ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ της υποστήριξης στο σύστημα εκπομπών, το ETS, όπως κάνετε εσείς κύριε Βάιμαν, και της επίδευξης στόχων οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή την μείωση της έντασης ενέργειας. Γιατί αν δεν δράσουμε όταν αλλάζουμε τους στόχους για την ε, ένταση ενέργειας και στο σύστημα ETS, ε έχουμε μία αντίφαση. <clears throat> Αν έχουμε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στην τιμή του άνθρακα και θα μειωθεί ακόμα περισσότερο η τιμή του άνθρακα, αυτό το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει. Ο κ. Κάρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία από τις σπάνιες ε, ενδιαφέρουσες συζητήσεις που είχαμε εδώ πέρα και ευχαριστώ τους δύο συγκητές μας, αλλά άκουσα κάποια πράγματα τα οποία είναι αξιοθαύμαστα. Ο κύριος Ζαντό είπε πως με την οικονομική ανάπτυξη θα ανέβουν οι τιμές του ρεύματος και θα γίνουν φτωχότεροι οι καταναλωτές. Αντιβαίνει τη λογική και την πείρα. Η ανάπτυξη σημαίνει ότι ο κόσμος έχει δουλειές και έχει μισθούς και άρα το ποσοστό του εισοδήματός τους που ξοδεύεται σε ενέργεια θα μειώνεται όσο αυξάνεται ο μισθός. Οπότε ο ένας μιλάει παράλληλα με τον άλλον, δεν ακούμε καθόλου και έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη των οικονομικών εδώ πέρα. Εξοικονόμηση έναντι της ε, κατανάλωσης, της έντασης ενέργειας. Έχουμε στόχο κατανάλωσης και στόχο έντασης. Στη χώρα μου τη Λετωνία οπωσδήποτε είμαστε πρωταθλητές στην εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι πολύ απλό μπορείτε να είστε πανφτωχοί. Όταν είστε πανφτωχοί συνεχώς εξοικονομείτε λεφτά. Δεν βλέπετε τηλεόραση γιατί κοστίζει. Κάθεσαι στο σκοτάδι και συζητάς και μιλά στην οικογένειά σου. φορά και το παλτό γιατί δεν ανάβεις τη θέρμανση, γιατί δεν έχει να πληρώσει. Οπότε, αν εστιάσουμε μόνο στόχους κατανάλωσης, αυτό το οποίο θα γίνει στη χώρα μου όταν αναπτυχθεί η οικονομία, είναι πως ο κόσμος θα χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια αποτελεσματι... ε, αναποτελεσματικά όπως έκαναν. Θα ξανανάψουν τις παλιές τις λάμπες, θα σπαταλάνε ενέργεια, αναφωτισμένο λεπτό ή όπως το μετράτε, θα ξανανοίξουν, θα ξαναβάλουν μπρος τα παλιά τους αυτοκίνητα που καίνε πολύ, θα ξανανοίξουν τα παλιά εργοστάσια που σπαταλάνε ενέργεια και ε, δημιουργούν ΑΕΠ αλλά σπαταλούν ε, ενέργεια. Οπότε αυτό το οποίο θέμε να κάνουμε είναι αυτό το οποίο κάνουν οι έξυπνες εταιρείε. Το έκανα και εγώ όταν ήμουν επιχειρηματίας. Εγώ κατασκεύαζα πάγο και πουλούσα στη Λετωνία και στη Φιλανδία. Ε, και εγώ εξοικονομούσα λεφτά με το να είναι όλη η εργασία χειροκίνητη. χρειάζεται περισσότερο πάγο, προσλαμβάνεις περισσότερους. Αλλά είναι σπατάλι. Πρώτα απ' όλα γιατί καμιά φορά δεν έρχονται οι άνθρωποι, αλλά κυρίω γιατί όταν κατασκευάζει κανεί με τα χέρια χρειάζεται πολύ χώρος για να αποθηκεύει τα αγαθά, γιατί δεν αποθηκεύει γρήγορα. Οπότε υπάρχει ψηλό κόστο ενέργεια, ηλεκτρισμού, γιατί χρειάζεται πολλά ψυγεία και μετά έλαβα την απόφαση, καθώς η εταιρεία μεγάλωνε και ήταν ασαφές το ποια θα ήταν η αγορά, επένδυσα σε αυτόματα μηχανήματα συσκευασία. Και βεβαίω κέρδισα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ε, τώρα ε, παράγω περισσότερα με μικρότερο κόστος. Και αυτομάτως και το περιθώριο κέρδους αυξήθηκε. Δεν χρειαζόμουν τόσο αποθηκευτικό χώρο. Έκανα παραγωγή σε μία μέρα με το κουμπί και κάνα δύο ανθρώπους αντί για 20 άτομα που να κάνουν τη δουλειά αυτή για 4-5 μέρες. Το ίδιο και σε μια οικονομία. Εντάξει, κοστίζει περισσότερο να είναι κανεί αποτελεσματικό, αλλά θέλουμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα έτσι ώστε όταν βγούμε από την κρίση θα έχουμε οικονομική ανάπτυξη με λιγότερη χρήση ενέργειας. Οπότε θέμε τους νέου λαμπτήρες, παραδείγματο χάρη, για να είναι πιο αποτελεσματική η βιομηχανία μα. Και θεωρώ άρα ότι εμεί που διαμορφώνουμε την πολιτική θα πρέπει να εστιάσουμε στο επίπεδο έντασης, γιατί ο μόνος τρόπος να μειωθεί τελικά η κατανάλωση είναι να φτωχύνει ο κόσμος, εάν δεν εστιαστούμε στην ένταση. Ε, αν δεν εστιαστούμε στην ένταση, είναι μείωση του πληθυσμού, η άλλη λύση, ή μεγαλύτερος πληθυσμός που θα ζει σε χαμηλότερο επίπεδο. Σκεφτείτε το δηλαδή. Ε, αν θέλετε να δείτε οικονομία, ελάτε στη χώρα μου, αλλά αυτό δεν είναι αποτελεσματικότητα ενώ ε, οργώνουν με, με το αλέτρι ακόμα. Και κόβουνε καυσόξυλα όπως έκαναν ε, πριν από αιώνε. Γιατί δεν, πήραν ποτέ, δεν αγόρασαν ποτέ αερόθερμο γιατί δεν είχαν λεφτά. Εντάξει, να έχουμε χαμηλή κατανάλωση ε, ε, αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, όχι επειδή είμαστε φτωχοί. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν την ένταση ενέργειας. Και μην ξεχνάτε, η Δανία διπλασίασε το ΑΕΠ χωρίς να αυξήσει την ε, παραγωγή ενέργειας. Οπότε είναι υπόδειγμα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 Πόσο, πόσο καιρό έχω 10 λεπτά, ναι. πόσο χρόνο έχω 10 λεπτά. Ακούσαμε πάρα πολλέ φιλοσοφικέ ε, ιδέε σε αυτή τη συζήτηση. Είναι πραγματικά συναρπαστική αυτή η συζήτηση. Λυπάμαι που ίσω δεν θα μπορέσω να δώσω απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Θα προσπαθήσω όμω να σταθώ σε ορισμένα σημεία. Από τη μία πλευρά το ερώτημα είναι ποιο είναι ο πραγματικό στόχο τη οδηγία. Και θέλω να τονίσω ότι δεν είναι ένας απόλυτος στόχος ο οποίος βασίζεται σε μια συγκεκριμένη βάση, αλλά αφορά μία αναφορά η οποία παρα... περιλαμβάνει και την αύξηση την οικονομική μέχρι το 2020 και επομένως είναι ουσιαστικά ένας στόχος έντασης εργασίας, ε, έντασης ενέργειας, συγγνώμη. Το δεύτερο ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσουμε και το οποίο περιλαμβάνω σε πολλές από τις παρατήρησεις των βουλευτών. Είναι καλό όταν σε φάσεις οικονομικής ε, ύφεσης ή χαμηλής ε, ε, ανάπτυξης να έχουμε ένα τέτοιο στόχο εξίσου καλό όπως σε εποχές οικονομικής ε, ανάπτυξης. Να σας πω εν συντομία την άποψή μου. Αυτό το οποίο είπε η κυρία Χόλ νομίζω ότι είναι πολύ σωστό και πολύ σημαντικό. Ότι ακόμα και σε περιόδους οικονομικής αδυναμίας είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρουμε και να προωθήσουμε μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Και συμφωνώ απόλυτα με τον Καρίν ότι το ερώτημα δεν είναι να βγούμε από την, <clears throat> από την ε, ύφεση, γιατί αν δεν έχουμε καταφέρει να περάσουμε κάποια μέτρα εξοικονόμησης, θα ανέβει πάρα πολύ γρήγορα η κατανάλωση ενέργειας. Πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι σε εποχή οικονομικής κρίσης θα έχουμε στο οικονομικό κύκλο, επομένω και λιγότερες επενδύσεις. Επομένω, αυτό κάνει πολύ δυσκολότερο να υπάρχουν οι αρχικές επενδύσεις, οι επενδύσει upfront, να χρηματοδοτηθούν στην αγορά. Και πρέπει να ζήσει κανείς και με αυτές τις πραγματικότητες. Θα πρέπει να προσπαθήσει φυσικά στο βαθμό του δυνατού να προχωρήσει ε, σε ανάπτυξη υπηρεσιών που θα βασίζονται στην εξοικονόμηση της ενέργειας, αλλά σε τελική ανάλυση, το ξέρουμε όλοι, οι αρχικές επενδύσεις είναι ένας παράγον τροχοπεδητικός και σε εποχές, της, ε, εποχές κρίσης δεν μπορούν εύκολα να γίνουν αυτές οι επενδύσεις παρά το γεγονός ότι σε τελική ανάλυση θα μπορούσαν να οδηγούσαν σε νέα ανάπτυξη και σε μεγάλες εξοικονομήσεις. Η τρίτη παρατήρηση που ήθελα εγώ να τονίσω είναι σε ένα ανώτερο κάπως υπέρτερο επίπεδο σε σχέση με την σύνδεση των διαφόρων εργαλείων, δηλαδή το θέμα του το εργαλείο της ε, ε, εμπορίας εκπομπών και της ε, χρήσης ανανεώσιμων ενεργειών και της ενεργειακής απόδοσης. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, επομένως δεν μπορώ να διεκδικήσω την η ικανότητα να κρίνω τα θέματα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί ε, εξέχοντες οικονομολόγοι όπως ο κύριο Στέρν ο οποίος τόνισε ότι πέραν των οικονομικών εργαλείων πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τη χρήση άλλων ενεργειών τα οποία υποστηρίζουν ή αντιτίθενται στις, στα οικονομικά μέτρα. Και η έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας ε, Ε, ε, ατομικής ενέργειας, ενέργειας ε, έδειξε ότι η χρήση πολλών εργαλείων δεν οδηγεί πάντα στον επιδιωκόμενο στόχο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο πρέπει να επιτύχουμε είναι να έχουμε μια ανάλυση επί τη βάση πολλών κριτηρίων. Θα πρέπει να λάβουμε τη δυναμική πτυχή, όχι μονάχα τα βραχυπρόθεσμα οικονομικά ε, ωφέλη που θέλει ενδεχομένως η αγορά να επιτύχει. Όλους αυτούς τους στόχους, τα πολλαπλά κριτήρια λοιπόν, δεν μπορούμε να τα επιτύχουμε <clears throat> με ένα μονάχα στόχο. Και αυτό το κάνει σαφές και η έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Ενεργείας. Αλλά ο κύριος Βάιμαν έχει δίκιο και αυτό φάνηκε και από διάφορα σχόλια. Άμα έχω πολλά εργαλεία, θα πρέπει να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός για την διάδραση μεταξύ όλων αυτών των ε, εργαλείων και μπορεί να είναι θετική η διάδραση αλλά μπορεί να είναι και αντίκη. Συζητήσαμε για το σύστημα εμπορίας εκπομπών αν παράλληλα με το σύστημα αυτό έχω πολιτικές προωθήσεις ε, ανανεώσιμης ενέργειας και εξοικονόμησης ε, ε, ενέργειας, θα πρέπει να σκεφτώ τι γίνεται με το όριο αυτό για τις εκπομπές, πώς θα πρέπει να τροποποιηθεί. Όταν λοιπόν έχουμε εργαλεία θα πρέπει να ξέρουμε πού είναι τα οικονομικά όρια και πού δεν είναι τα οικονομικά όρια. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε συζητήσει σε βάθος και θα πρέπει να συλλέξουμε και εμπειρικά στοιχεία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη σκέψη μας. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο είναι σημαντικό και στην ε, οδηγία ότι είναι τα μέτρα τα πρέπει να έλκονται από τη στοχοθεσία. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και ποιο είναι το μήνυμα το οποίο έρχεται από τους στόχους. Η συζήτηση τώρα για το αν είναι καλύτερη η διατύπωση με απόλυτους στόχους ή με ένταση ενέργειας δεν θα λάβω θέση στο θέμα αυτό, αλλά είναι σαφές ότι ο τρόπος με τον οποίο, έχει, με τον οποίο παρουσιάζεται ο στόχος πρέπει να δώσει ένα σημαντικό μήνυμα και έχει μεγάλη σημασία και η ψυχολογική, ο ψυχολογικός αντίκτυπος ενός στόχου από την οικονομική σημασία του στόχου. Θα περιοριστώ λοιπόν σε αυτά τα σχόλια που θέλω να κάνω. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να σχολιάσει κανείς. Αλλά θα ήθελα εν κατακλείδη να πω ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν θέτουμε ένα στόχο να σκεφτούμε και την εποπτεία, την παρακολούθηση της επίτευξης αυτού του στόχου. Έχουμε συζητήσει σε μεγάλο βαθμό και το θέμα της ε, οδηγίας για τις υπηρεσίες και την επίπτωση της ενέργειας στον τομέα αυτό. Όλοι μας ε, πιστεύω οι περισσότεροι από εμά έχουν κάνει πανεπιστημιακές σπουδές, αλλά όταν ασχολείται κανείς με τα θέματα σε καθημερινό επίπεδο, πολλές φορές νιώθει σύγχυση με τον τρόπο με τον οποίο ε, διατυπώνται αυτά τα πράγματα, πώς θα συνδυαστεί δηλαδή ένας απόλυτος στόχος μείωσης ή ένας σχετικός ε, στόχος με την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Θα ήθελα λοιπόν να επιχειρηματολογήσω υπέρ του να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι να τον ε, διάφανο και ευνόητο. Ευχαριστώ ο καθηγητής Βάιμαν. Ναι. Έγιναν πολλές παρατηρήσεις. Θα ξεκινήσω με την κυρία Χολ. Με τη δική της ε, παρέμβαση είπε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πως εάν εξοικονομούμε ενέργεια δεν είναι κόστος. Αυτό είναι καινοτομία. Δυστυχώ δεν ισχύει αυτό. Όταν εξοικονομούμε ενέργεια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πόρους. Εάν θέλουμε να κάνουμε ένα καλύτερο ψυγείο, θέλουμε να το μονώσουμε καλύτερα. Αυτό κοστίζει περισσότερο από ένα λιγότερο μονομένο ψυγείο. Το ίδιο και για ένα σπίτι. Που είναι πολύ ακριβή μόνωση σε ένα σπίτι. Εάν έχουμε ένα κτίσμα του 1970 και θέλουμε να το φέρουμε στην κατάσταση ενός νέου κτίσματος, μιλάμε για 50 έως 80 ευρώ σε τέτοια μέτρα μόνωσης. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη αυτό το κόστος όταν σκεφτόμαστε το που μπορούμε καλύτερα να εξοικονομήσουμε. Το να το αγνοούμε είναι παράλογο. Και επιτρέψατε μου να κάνω μια παρατήρηση στον Πρωθυπουργό σας εγώ θα συνιστούσα να αλλάξει συμβούλους ενέργειας. Η παρατήρηση ότι ποτέ μια αγορά δεν τήρησε προθεσμία ε, δεν ισχύει όσον αφορά το ε, εμπόριο εκπομπών. Πώς λειτουργεί το εμπόριο εκπομπών. Ορίζουμε ε, ένα πλαφόν και αυτό λειτουργεί από την πρώτη μέρα στην Ευρώπη ως επιχείρηση μπορεί κανείς να εκπέμψει εάν έχει μόνο μία άδεια. Και η ποσότητα για την οποία υπάρχουν άδειες είναι περιορισμένη και αυτό ισχύει από την πρώτη μέρα. Δεν υπάρχει προθεσμία. Και αγορά λειτουργεί θαυμάσια. Έχουμε τα μηνύματα, βεβαίως εντάξει τα μηνύματα των τιμών δεν είναι αυτά τα οποία χρειαζόμαστε λέει η αγορά. Α, αυτά τα οποία κάνει η πολιτική. Ο Πρωθυπουργό λοιπόν θα έπρεπε να τα σκεφτεί αυτά την επόμενη φορά που θα ρωτήσει τους ειδικού του. Δεύτερη απάντηση στον κύριο Τούρμες. Με παρεξηγήσατε. Εγώ δεν είπα πως ε, πρέπει να κάνουμε την πολιτική που κάνουμε τώρα και μετά να προσαρμόσουμε ε, το πλαφόν. Είπα πως πρέπει να προσαρμόσουμε το πλαφόν και μετά να μην κάνουμε τίποτα άλλο. Και να αιτιολογήσω γιατί. Το εμπόριο εκπομπών λειτουργεί με βάση μια αρχή. Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο να αρέσει στους οικονομολόγους η αρχή είναι η εξή. Όρισε το πλαφόν, όρισε τον πολιτικό στόχο και μετά κάνει αυτό το στόχο δεσμευτικό με το να δώσει δικαιώματα και να λες όποιος έχει αυτό το δικαίωμα επιτρέπεται μόνο να επιβαρύνει το περιβάλλον μας. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πώς επιτυγχάνω την τήρηση αυτού του πλαφών. Και η απόφαση αυτή που με ποιο μέσο, ποια τεχνολογία κτλ. αποφεύγουμε, θα το αποφασίσει το σύστημα αυτό εμπορές εκπομπών με το να δρουν αποκεντρωμένα οι επιχειρήσει και με καλό λόγο. Γιατί, γιατί πρώτον αυτοί έχουν τις πληροφορίες που χρειάζεται για να διαπιστώσουν πού τελικά είναι πιο φτηνό να γίνει αυτό και μέσω του εμπορίου έχουν το κίνητρο ακριβώς να εκμεταλλευτούν αυτές τις πληροφορίες. Είναι λοιπόν προς το συμφέρον μιας επιχείρησης να ψάξει πού μπορώ να εξοικονομήσω με τον καλύτερο τρόπο διοξιδίου του άνθρακα για να πουλήσω μετά τα δικαιώματα και να κερδίσω λεφτά. Το μέσο αυτό είναι αυτό το οποίο λένε οι οικονομολόγοι ένα κίνητρο, είναι προς το συμφέρον ε, των ανθρώπων αυτών. Γι' αυτό λειτουργεί καλά. Γι' αυτό δεν έχουμε ε, κάποια μέσα ελέγχου. Εάν το γυρίσουμε ανάποδα, το αντιστρέψουμε και πούμε θα έχετε αυτή η χύψη και τη ψή τεχνολογία, τι κάνουμε, μειώνουμε το πλαφόν γιατί έτσι έχουμε θέση εκτός το εμπόριο εκπομπών με, όλες του, με όλη του την ισχύ γιατί ε, λένε μπορούμε να μειώσουμε το πλαφόν και τα λοιπά, αλλά είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν αντιλαμβάνεται το πώς λειτουργεί ο, η αγορά αυτή. Επιτρέψατε μου ε, μία τελευταία παρατήρηση. Να πούμε κάτι απλό. Δηλαδή, η Κομισιόν θα μπορούσε η Κομισιόν να θέσει κατευθείαν το στόχο στο 30%. Ναι, κοιτάξτε, το πώς, το πώς, μια που μιλάμε για το πλαφόν, το πώς θα το επιλέξουμε αυτό είναι μια πολιτική απόφαση των πολιτικών. Εδώ, στις Βρυξέλλες θα το διαπραγματευτείτε, δεν είναι η δικιά μου δουλειά να το ορίσω ως οικονομολόγος. Το δικό μας το μήνυμα είναι, αν θέλουμε να αποφύγουμε το διοξείδιο του άνθρακα, προσωπικά εγώ θεωρώ πως πρέπει να το κάνουμε, τότε είναι μια λογική ιδέα να γίνει με αποτελεσματικότητα κόστους. Τώρα αν είναι 10, 20, 30 ή 40% ναι. Αλλά όποιο και αν είναι αυτό το ποσοστό είναι πολιτική απόφαση που πρέπει να ληφθεί με μια δημοκρατική διαδικασία. Τώρα. Έχω ακόμη πέντε λεπτά, ε. Τώρα, ε, μιλήσαμε για μια έτσι φιλοσοφική συζήτηση. Α, εγώ θεωρώ ότι ήταν οικονομική παρά φιλοσοφική. Επιτρέψατε μου να αναφέρω μια τελευταία θεμελιώδη παρατήρηση. Αυτό το οποίο παρατήρησα συζήτηση είναι πως προφανώς υπάρχει διαδεδομένη άποψη πως η εξοικονόμηση ενέργειας είναι αυτής ένας καλός στόχος, κάτι το οποίο ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι. Έχουν δύο επιχειρήματα. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο είπατε. Πράγματι η κατανάλωση της ενέργειας από μόνη της δεν είναι κάτι το κακό. Εμείς χρησιμοποιούμε ενέργεια και αυτό είναι σωστό γιατί μπορούμε να κοιταζόμαστε τώρα και να μιλάμε στο μικρόφωνο και να ακουγόμαστε. Χρησιμοποιούμε ενέργεια με λογικό τρόπο. Ε, εγώ θα ήθελα να φέρω ένα άλλο επιχείρημα. Ε, να κάνουμε ένα πείραμα, σκεφτείτε. Φανταστείτε πως είχαμε μια πηγή ενέργεια στην Ευρώπη, η οποία είναι ανεξάντλητη, δεν βλάπτει το περιβάλλον, τελείως καθαρή ας πούμε, μια ουτοπία έτσι, σκεφτείτε το. Και και απολύτως καθαρή και ανεξάντλητη, τίποτα, τίποτα, κανένα πρόβλημα περιβαλλοντικό και μπορεί να παρεχθεί με κάποιο μέσο κόστος. Θα καθόμαστε να μιλάμε για αυτή την οδηγία εξοικονόμησης ενέργειας. Όχι! Μιλάμε γι' αυτό γιατί με τη χρήση της ενέργειας έχουμε την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και το ότι δεν είναι ανεξάρτητοι πόρη. Αυτά είναι τα προβλήματα. Εάν έχουμε λοιπόν στόχους πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά τα ουσιαστικά προβλήματα. Αλλά το να λέμε πρέπει να εξοικονομήσουμε ενέργεια από μόνο του ε, δεν είναι παράλογο, ε, δεν είναι λογικό. Είναι παράλογο αν με ρωτήσετε. Εάν δεν επικεντρωθούμε σε αυτούς τους στόχους. Εάν το κάνετε αυτό θα λύσετε πολλά προβλήματά σας και τα πολλά προβλήματα που ανέφερε ο κύριο Άιχαμερ. Γιατί πολλά από τα περίπλοκα προβλήματα εδώ πέρα προκύπτουν από το ότι υπάρχουν διαφορετικοί στόχοι. 20% εξοικονόμηση της ενέργειας, 20% περισσότερη αποτελεσματικότητα, 20% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα και δεν έχουμε σχέδιο για το πώς θα γίνει αυτό. Όχι, όχι, δεν, δεν υπάρχει. Ε, είναι σαφές από αυτή τη συζήτηση. Και θεωρώ πως πρέπει να συζητήσουμε το πραγματικό πρόβλημα. Και το πραγματικό πρόβλημα, κατά την άποψή μου, είναι το πρόβλημα του κλίματος και το πρόβλημα των πόρων. Αλλά όχι αφ' η κατανάλωση της ενέργειας. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Και μια ε, παρατήρηση για τον συνάδελφο εγώ είμαι, συμφωνώ μαζί σας πως πρέπει να συζητήσουμε το πώς ε, τα διάφορα μέσα συνδυάζονται, αλλά ε, αυτό το οποίο με ενοχλεί εμένα σε αυτό είναι πως τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται για να αιτιολογήσουν γιατί ε, επαρκεί το εμπόριο εκπομπών δεν συζητούνται πραγματικά. Δεν συζητείται το ζήτημα του κόστους. Δυστυχώς δεν υπάρχουν όλα αυτά συζήτηση. Αυτά. Και νομίζω πως ε, τελείωσα και πιο νωρί. Μάλιστα σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους κυρίους Άχερμαν και Βάιτμαν. Βάιτμαν. Μάλιστα. Τον καθηγητή κύριο Βάιμαν και τον δόκτωρα Άχερμαν. Νομίζω πως ήταν ε, άξιζε ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Okay. Einverstanden. Meine Damen und Herren, wir fahren. Μάλιστα, συμφωνώ. Συνεχίζουμε κυρίε και κύριοι. Έχουμε ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη ακόμα. Ich, äh, δηλαδή το σημείο 5. Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Στον τομέα της ενέργειας έχουμε τον αγαπητό συνάδελφο Κάρινς, τον εισηγητή πρώτα απ' όλα. Ε, δεν ξεκινάμε αν δεν αφήσετε τον κύριο Κάρινς να μιλήσει. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Είμαστε όλοι λίγο κουρασμένοι, λέει ο κ. Κάριν. Συζητάμε για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί τη βάση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου τον Φεβρουάριο για τις συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τρίτες χώρες στον τομέα της ενέργειας. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει και τα στοιχεία να κυκλοφορούν έτσι ώστε να επιλέγονται οι βέλτιστες πρακτικές και να πλησιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια κοινή φωνή θα λέγαμε και κοινή θέση απέναντι στους παροχείς εισάγουμε το 80% του πετρελαίου, το 60% του φυσικού αερίου, Τα ποσοστά αυτά δυστυχώς αυξάνονται και δεν μειώνονται. Και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο η Ρωσία είναι ένας από τους βασικούς προμηθευτές, είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής για το αέριο και σχεδόν ο μεγαλύτερος στο πετρέλαιο όπως και οι χώρες ΟΠΕΚ Επίσης και η Νορβηγία είναι μεγάλος προμηθευτής. Υπάρχουν 60 διακυβερνητικές συμφωνίες για το φυσικό αέριο και 30 διακυβερνητικές συμφωνίες για το πετυρέλαιο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη για, την, για τις σωστές πρακτικές οι οποίες ακολουθούνται. Η Ρωσία γνωρίζει σαν παράδειγμα το περιεχόμενο όλων των συμφωνιών που έχουμε συνάψει με τη Ρωσία. Αλλά δεν γνωρίζουμε εμείς το αντίθετο. Μία χώρα δεν γνωρίζει τις συμφωνίες της Ρωσίας με τις άλλες χώρες. Είναι μονόδρομος. Γνωρίζουν τα πάντα για μας, αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε ακριβώς το τι ρήτρε, τι πρακτικές και τι συμφωνίες έχουν γίνει. Η ανησυχία από πλευράς Ευρωπαϊκής λοιπόν είναι αν ο νόμος επιτρέπει να δοθούν εγγυήσει για τις εισαγωγές αυτές ή αν θα πρέπει οι διακυβερνητικές συμφωνίες να είναι αυτές οι οποίες παρέχουν τις αντίστοιχες εγγυήσει. Μια χώρα ας πούμε που θέλει να δημιουργήσει νέες υποδομές και υπάρχει μια συμφωνία με τη Ρωσία, η Ρωσία η οποία θέλει να πιέσει προς την κατεύθυνση αυτή τις πληροφορίες που θέλει για να πιέσει και τρίτες χώρες. Και μια τέτοια συμφωνία υπογραφή με πίεση της Ρωσίας, τότε σε αυτήν την περίπτωση η επένδυση θα κοστίζει όλο και περισσότερο, θα, τεθεί, θα, τεθούν, θα δημιουργηθούν πολλά ερωτηματικά σε σχέση με τον στόχο της συγκεκριμένης υποδομής και όλα αυτά θα δημιουργήσουν υπερβολικό κόστος και προσδοκίες. Νομίζω λοιπόν ότι το κίνητρο που δίδεται τώρα είναι ένα καλό κίνητρο. Νομίζω ότι θα πρέπει σαν βουλευτές να υποστηρίξουν την πρόταση. Υπάρχουν ανησυχίες ανάμεσα σε ορισμένα κράτη-μέλη για θέματα κυριαρχίας. Πολλές χώρες αναρωτιούνται αν θα ανακατεύονται οι Βρυξέλλες περισσότερο στα θέματα τους. Υπάρχουν προβλήματα και στις βιομηχανίες σχετικά με τις ρήτρε εμπιστευτικότητας. Από ό,τι φαίνεται το θέμα της εμπιστευτικότητας όμως καλύπτεται γιατί η νομοθετική ρύθμιση αυτή που προτείνεται ασχολείται με τις διακυβερνητικές συμφωνίες και όχι με τις συμφωνίες ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία λοιπόν υπάρχει μια ξεκάθαρη αναφορά στην εμπορική συμφωνία, η οποία απαιτείται να γνωστοποιηθεί, και μόνο στην προτινόμενη ε, νομοθεσία οι χώρες μπορεί να απαιτήσουν όρους εμπιστευτικότητας για το σύνολο της συμφωνίας. Οπότε θα γνωρίζει έτσι κι αλλιώς τότε ποιο είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν γίνεται ή δεν γίνεται σεβαστός ο κοινοτικό νόμος. Αλλά τώρα εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες για τιμολογήσεις, για μεγέθη κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα κρατούν τα κράτη-μέλη. Η εμπιστευτικότητα λοιπόν ως προς το προτινόμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι πρόβλημα. Αν διαβάσουν σωστά την πρόταση και αν εμείς δεν στρεβλώσουμε την ισορροπία με δεν θα επηρεαστεί το θέμα της εμπιστευτικότητας και τα επαγγελματικά ε, απόρριτα δεν θα δημοσιοποιηθούν. Ένα άλλο εμπόδιο το οποίο θα έχουμε είναι θεσμικού τύπου. Οι αρμοδιότητες των κρατών μελών από τη μία με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την άλλη θα έρθουν σε αντιπαράθεση. Εδώ σαν βουλευτές και σαν προασπιστές της ιδέας μιας κοινή αγοράς και στον τομέα της ενέργειας, νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις, γιατί είναι το πρώτο νομοθετικό βήμα το οποίο μας οδηγεί ε, προς μια κοινή ενεργειακή πολιτική προς μια κοινή αγορά ενέργειας. Είμαστε μακράν βέβαια ακόμα, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω λοιπόν ότι αν σταθμίσουμε σωστά τα ωφέλη και το κόστος, τότε θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε σωστά και τις δυνατότητες που έχουμε για τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες όπως η Ρωσία και να σταθμίσουμε το κόστος αυτών των συμφωνιών ιδιαίτερα για χώρες οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα αυτόνομες στον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύονται. Πρέπει να το ζητήσουμε αυτό λοιπόν από τα κράτη-μέλη, γιατί όπως είπα ως προς το επαγγελματικό απόρριτο δεν υπάρχει πρόβλημα. Και κλείνοντας, υπάρχουν ορισμένα άρθρα στα οποία νομίζω μπορούν να υπάρξουν τροπολογίες για βελτιώσεις, αλλά νομίζω ότι οι βασικές γραμμές της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι, πρέπει να υποστηριχθούν μας οδηγούν πιο κοντά σε μια ενεργειακή κοινή αγορά και μια κοινή φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν διαπραγματεύεται και συζητά με τους ιδιοκτήτες σε εισαγωγικά των πηγών ενέργειας. Ο κύριος Γκλάντε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δυστυχώς λείπουν κάποιοι συνάδελφοι και θέλω να εκπροσωπήσω τον κύριο Λάγκε, ο οποίος έχει την εξής άποψη. Θεωρεί ότι είναι μια σωστή πρόταση και μέσα από την ε, νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας θα πρέπει να υπάρξει μια συνένωση συμβερόντων και τα θέματα αυτά. Παραγωγικά χάρη συμφωνίες όπως αυτή με την ε, Νορβηγία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει να υπάρξει μια, ένα συντονισμό των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια κοινή εμπορική στάση προς τα έξω. Ο κ. Λάγκεν ζητάει στο άρθρο 5 να υπάρξει μια δυνατότητα επαλήθευσης στο άρθρο 6 δεν είναι σαφές πώς θα γίνει ο συνδυασμός των διαφόρων πηγών ενέργειας. Χρειαζόμαστε σαφείς ε, προδιαγραφές. Ένα άλλο σημείο αφορά την ε, απόρριψη της ε, ανοιχτής μεθόδου συνεργασίας για τα θέματα αυτά. Εγώ θέλω απλώς να να πω κάτι από τη δική μου πλευρά, εφόσον έχω το μικρόφωνο, είπε ο εισηγητή προηγουμένω. Υπάρχει η ανάγκη πληροφόρηση της Κομισιόν, ανακοίνωση στην Κομισιόν, μόνο για διακρατικές συμφωνίες. Θα ήθελα να ξέρω όμω ποια είναι η ισορροπία μεταξύ των διακρατικών συμφωνιών με τις ιδιωτικές συμφωνίες. Γιατί στη δική μου χώρα τουλάχιστον είναι περισσότερες, είναι σχεδόν αποκλειστικά ιδιωτικές συμφωνίες, δεν γίνονται διακρατικές συμφωνίες που να εμπλέκουν τη Γερμανία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζαντός Σκιώδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα δείτε ότι μπορώ να συμφωνώ και με τον κύριο Κάριντς από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανάμιξη μεταξύ στόχων και μέσων. Οι πρώτες της Κομισιόν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι σαφές αυτό ότι θέλουμε να έχουμε ένα πιο έντονο συντονισμό μεταξύ των δράσεων των κρατών μελών και με τις, των εσωτερικών νομοθεσιών τους στον τομέα της ενέργειας. Θα υποστηρίξουμε λοιπόν και εμείς τον εισηγητή, ο οποίος από τη δική του πλευρά υποστηρίζει την κίνηση της Κομισιόν εγώ είμαι συντάκτης γνωμοδότησης στην Επιτροπή ε, Εξωτερικού Εμπορίου. Στο σημείο 5, στο άρθρο 5 που αφορά τον έλεγχο εκ των προτέρων, θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο, ο έλεγχος της Κομισιόν και να έχει ένα χαρακτήρα αυτεπάγγελτο και αυτόματο και όχι να έχει μια εθελοντική μονάχα μορφή από την πλευρά της Κομισιόν. Για το άρθρο 3 που αφορά τις υφιστάμενες συμφωνίες, συμφωνίες που είναι υποδιαπραγμάτευση, θεωρούμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητήσει από το αντίστοιχο κράτος μέλος να υπάρξει μια επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας όταν έρχεται σε σύγκρουση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή τους ευρωπαϊκούς στόχους σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά θέματα. Αυτό το είπε και ο ίδιος ο κύριος Κάρινς, το υπενθύμησε. Δεν πρέπει να έχουμε σύγχυση η οποία οδηγεί σε αμφισημίες και βαραίνει τη συζήτησή μας για το θέμα των διακρατικών συμφωνιών και των εμπορικού χαρακτήρα ιδιωτικών συμφωνιών. Εγώ νομίζω πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη, μεγαλύτερη διαφάνεια για τα θέματα αυτά και αυτό θα μας επιτρέψει να μην περάσουμε σε συζητήσεις οι οποίες δεν έχουν και ιδιαίτερο νόημα. Επίσης, για το θέμα των ε, ε, εξαιρέσεων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε τρίτους και σε ενεργειακές ε, δομές και εδώ πρέπει να υπάρχει μια κοινοποίηση της άρνησης για την πρόσβαση τρίτων στις ενεργειακές μας υποδομές. Αυτό έχει να κάνει με τα θέματα ενεργειακής ασφάλειας και διαφάνειας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά <clears throat> για να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε υποδομές οι οποίες δεν θα χρησιμοποιηθούν πλήρως. Τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω. Θα πρέπει στη συζήτηση αυτή να προσθέσουμε και ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο εγγράφεται αυτή η συζήτηση. Συζητούμε ήδη για τον οδικό χάρτη του 2050 και συγχρόνως για τους κλιματικούς στόχους, τους στόχους ενεργειακής ασφάλειας. Νομίζω ότι και σε αυτήν την περίπτωση οι σκέψεις μας σε σχέση με τις διακρατικού χαρακτήρα αυτές συμφωνίες και των υποδομών που προέρχονται από αυτές τις συμφωνίες θα πρέπει όλα αυτά να εγγραφούν σε μία προοπτική μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης και μείωσης εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου που να είναι συμβατές αυτές οι ενέργειες λοιπόν και με την ενεργειακή νομοθεσία της Ευρώπης. Λοιπόν, μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια, μεγαλύτερη βιωσιμότητα και αηφορία. Νομίζω ότι είναι οι στόχοι τους οποίους θα πρέπει να θέσει η Επιτροπή μας ενισχύοντας την σωστή κατεύθυνση των προτάσεων της Επιτροπής. Ο κ. Μπαλτσίτης. E, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον συνάδελφο για το έγγραφο το οποίο μας παρουσίασε, σημαντικό έγγραφο, διδιεγγυήσεις στην ανάπτυξη της αγοράς και μειώνει την πολιτική πίεση προς κάποια κράτη-μέλη, πίεση που δημιουργείται από την εισαγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου. Αυτά τα έχει πει και τα απασχολούν και τον Επίτροπο Έτιγκερ, ο οποίο πιστεύει ότι μόνο μία πραγματικά ενιαία αγορά μπορεί να διασφαλίσει την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Η αξιολόγηση βέβαια της διαδικασίας αυτής γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Ξέρετε ότι τεράστιες επενδύσεις, εκατομμύρια επενδύσεις χρειάζονται Πρέπει να δημιουργηθούν τα απαιτούμενα δίκτυα, πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές. Δεν είναι καθόλου εύκολο να εφαρμόσει κανείς το σχέδιο το οποίο έχει. Αυτό οφείλεται στο ότι ε, νιώθουμε έντονα την πολιτική πίεση η οποία ασκείται. Υπάρχουν πολλοί πολιτικοί οι οποίοι θέλουν να παρεμποδίσουν την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων τα οποία προτείνουμε εμείς. Θα πρέπει να κατανοήσουμε επίσης ότι η συγκεκριμένη πίεση παρεμποδίζει τις επενδύσεις από πλευράς ορισμένων ανασφαλών επενδυτών και με αμφισβητούμενη ε, επιτυχία των επενδύσεών τους. Αυτό το είδαμε και στο βορρά της Ευρώπης με τον αγωγό Nord Stream υπήρξαν ορισμένοι ηγέτες που πιστεύουν ότι το τρίτο πακέτο θα πρέπει να αναθεωρηθεί έτσι ώστε να γίνει πιο κατανοητό για τις τρίτες χώρες. Αυτό σημαίνει στην ουσία ότι θα πρέπει να γίνει πιο ουδέτερο. Κάτι τέτοιο μας ανησυχεί για το πόσο είναι εφικτή η πολιτική που θέλουμε να εφαρμόσουμε στο μέλλον. Νομίζω ότι η διαφάνεια του συγκεκριμένου εγγράφου, κειμένου, είναι κάτι το οποίο δεν δημιουργεί αμφιβολίες. Πρέπει να βελτιώσουμε την προστασία, την προστασία των αγορών μας και αυτό θα το πετύχουμε με διάφορα μέσα. Υπάρχει ένα θέμα όμως εδώ, ο καθορισμός των τιμών. Όταν μιλάμε για ανταλλαγή πληροφοριών, και αν τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν, ε, μεσολαβητή με τις τρίτες χώρες, τότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό καθορισμού των τιμών. Ξέρουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο καθορίζονται οι τιμές διαφέρει από τόπο σε τόπο και νομίζω ότι το συγκεκριμένο έγγραφο θα μας βοηθήσει στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Πάντως κατά τα άλλα έχει σημασία η πρόταση αυτή και είναι κάτι το οποίο θα βελτιώσει την αγορά στο μέλλον. Ο Βιντάλ Κουάντρας. Ο κύριος Βιντάλ Κουάντρας, ευχαριστώ πρόεδρε. Η πρόταση αυτή απόφασης είναι παράλληλη με την ανακοίνωση της Κομισιόν σε σχέση με την ασφάλεια εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία που συζητούσαμε πρόσφατα. Και εγγράφεται σε ένα γενικότερο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει σαν στόχο από τη μία πλευρά να είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος και συγχρόνως ο καθένα θέλει στο ίδιο σκάφος να κάνει του κεφαλιού του. Αυτά όμως δεν μπορούν να γίνονται στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να έχει ο καθένας τη δική του δημοσιονομική πολιτική, ενώ έχουμε μια ενιαία νομισματική πολιτική. Όλα αυτά μας οδηγούν σε μια καταστροφή. Θέλουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας, αυτό είναι πολύ καλό για όλους. Από την άλλη πλευρά λέμε ότι ο καθένας έχει τη δική του κυριαρχία για το ενεργειακό του μείγμα, για να συνάπτει συμφωνίες διμερείς και διεθνείς για την τροφοδοσία ενέργειας, όπως θέλει. Και αυτό φυσικά θα μας οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα αν παίρνει ο ένας αποφάσεις μονομερείς για το μίξ, για το μήμα. Αυτό έχει προφανείς οικονομικές συνέπειες για όλους. Εάν λοιπόν υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες οι οποίες είναι διμερούς χαρακτήρα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι επιπτώσεις του γιατί κάποιες από τις ρήτρες τους έμεσα ή άμεσα επηρεάζουν και άλλα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί λοιπόν η κοινότητα να μιλάει με, η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάει μονάχα με μία φωνή. Γι' αυτό πιστεύω ότι όπως είπε ο συνάδελφος Κάρινς αυτή η πρόταση δεν περιορίζει την κυριαρχικότητα των κρατών μελών, απλώς εισάγει ένα μηχανισμό που είναι η παρουσία της Κομισιόν ως παρατηρητού, εάν θέλει, εάν ή αλλιώς θα το ζητήσει κάποιο κράτος μέλος, να είναι παρατηρήτρια η Κομισιόν στη διαδικασία ε, διαπραγματεύσεων και στη συνέχεια θα εκφραστεί εξάντε για την σκοπιμότητα αυτής της συμφωνίας. Όλα αυτά δεν εμποδίζουν ένα κράτος να προχωρήσει σε μια διμερή συμφωνία, αλλά τουλάχιστον θέτει κάποια περιοριστικά όρια, κάποια, κάποιους φραγμούς για να αποφύγει ότι μια τέτοια συμφωνία θα είναι βλάβερη για άλλα κράτη-μέλη και έτσι ότι θα βλάπτει και θα παραβιάσει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Σύμφωνο λοιπόν με τον Κάρενς και με τον Ζαντό σε κάποιο βαθμό ότι αυτή η πρόταση πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. την εμπιστευτικότητα νομίζω ότι δίνει τις κατάλληλες εγγυήσει ώστε να μην υπάρχει καμία ανησυχία. Κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα. Ε, Ευχαριστώ. Εγώ στηρίζω το έγγραφο, θεωρώ πως είναι σημαντικό να συμφωνούμε όλοι. Θέλω να πω κάτι, φοβούμαι πως οι συνάδελφοι, τα κράτη-μέλη, θα το εξασθενήσουν αυτό εδώ πέρα στο Συμβούλιο, γιατί κανείς δεν θέλει να δίνει πληροφορίες, να τον ελέγχουν οι άλλοι κτλ. Οπότε πρέπει να δώσουμε μία μάχη για να μην συμβεί αυτό. Δεύτερον, επειδή κανείς δεν θέλει να δίνει πληροφορίες, βεβαίως πληροφορίες είναι κάποια δύναμη, κάποια κυριαρχία, εξουσία κτλ. Θεωρώ πως ο αριθμός ε, των ε, διακρατικών συμφωνιών θα μειωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί θα τις λένε εμπορικές συμφωνίες π.χ. Nord Stream. Δεν είναι διακρατική συμφωνία, είναι εμπορική συμφωνία. Οπότε τι θα γίνει, θα παρακάμψουν το θέμα. Οπότε σκέφτομαι πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε. Εάν μπορούμε, έτσι. Τι μπορούμε να βάλουμε στην έκθεση για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Το θέμα ατόπιν αφορά τον ορισμό της ακρατικής συμφωνίας. Ε, αν υπάρχουν κάποιοι όροι, κάποια γνωρίσματα με τα οποία εμείς τα λέμε είναι η συμφωνία διακρατική. Ευχαριστώ πολύ. Εάν μου επιτρέπετε συνάδελφοι έχουμε ε, κάποιους προσκεκλημένους από την ΕΟΚΕ στους οποίους θα ήθελα να δώσω το λόγο. Εάν θέλετε μπορείτε να, να μιλήσετε για λίγα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Η ΕΟΚΕ προετοιμάζει τη σχετική της γνωμοδότηση που ελπίζουμε να περάσει από την Ολομέλειά μας στα μέσα Ιανουαρίου. Ήδη συνεδρίασε η ομάδα μελέτης, ο εισηγητής υποστηρίζεται από μια ομάδα ε, μελέτης και μετά πάει στην Επιτροπή, στο τμήμα όπως το λέμε και μετά στην Ολομέλεια. Οπότε οτιδήποτε σας πω σήμερα είναι προσωπική άποψη αν και βασίζομαι σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις, αλλά ακόμα δεν έχει εγκριθεί ακόμα η γνωμοδότησή μας. Οπωσδήποτε καλωσορίζουμε την προτινόμενη απόφαση, νομίζουμε πως, σύμφωνα με το άρθρο 194 της συνθήκης με την ενεργειακή στρατηγική για το 2020 και πολύ έχουμε αργήσει κιόλα. Επίσης καλωσορίζουμε το ότι θα απαιτείται πληροφορίες ε, θα απαιτούνται πληροφορίες για όλες τις υφιστάμενες συμφωνίες και απορούμε που δεν έχει γίνει ήδη κάτι τέτοιο. Θεωρούμε εδώ πέρα πως πρέπει να γίνει μια πρόβλεψη για την εμπιστευτικότητα. Άκουσα αυτά τα οποία είπε ε, εισηγήτρια και άλλοι και λέει πως δεν είναι ζήτημα η εμπιστευτικότητα. Εμεί θεωρούμε πω είναι ζήτημα, αλλιώ θα είχε ήδη υπάρξει μια τέτοια συμφωνία. Και οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ενωμένη φωνή. Καλωσορίζουμε το άρθρο 5, όπου θα πρέπει να υπάρχει μια επίσημη δήλωση της Κομισιόν για την συμβατότητα, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι για το χρόνο αυτό των τεσσάρων μηνών, στον οποίο μετά η, συμφων... η σιωπή θεωρείται συνένεση. Εμείς θα θέλαμε μια επίσημη συνένεση. Επίσης ανησυχούμε για τον αποκλεισμό εμπορικών συμφωνιών, ειδικά όπου εμπελέκονται ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές. Βεβαίω εδώ πέρα και αν έχει ρόλο η εμπιστευτικότητα, αλλά οι καταναλωτές δεν θα χαρούν με τη διάκριση αυτή που κάνουμε. Επίσης, απορούμε πως δεν έχει γίνει πλήρης ακόμα μελέτη επιπτώσεων, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα, όπως υπόθηκε, για τα κράτη-μέλη και μπορεί να θεωρήσουν πως ε, υπάρχουν κάποιες αρμοδιότητες που μεταφέρονται εδώ πέρα από το παράθυρο. Και τέλος ε, θα πρέπει να γίνει διάμεση αξιολόγηση μετά από δύο χρόνια και όχι τέσσερα. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε με το νέο έτος να μοιραστούμε μαζί σας την τελευταία μας αξιολόγηση. Κύριε Ζήλα λοιπόν από την Κομισιόν, αν θέλετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ. Να ευχαριστήσω επίσης και για τις προτάσεις που έγιναν για βελτίωση και ενίσχυση του κειμένου. Ένα θέμα μόνο Ο στόχος μας είναι και μια μεγαλύτερη διαφάνεια ανάμεσα στα κράτη-μέλη και η ανάγκη να υπάρξει ένα αξιόπιστο σύστημα το οποίο να επιτρέπει στα κράτη-μέλη να μοιράζονται τις πληροφορίες μεταξύ τους και όχι μόνο όταν οι συμφωνίες αυτές δημοσιεύονται. Να υπάρξει ένας μηχανισμός δηλαδή μέσω του οποίου τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να αυξήσουν την διαφάνεια των στοιχείων τους και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε τη συμβατότητα των συμφωνιών αυτών με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στον τομέα της ενέργειας. Είναι μια νομοθεσία η οποία διευρύνεται και η οποία θα έλεγα αφορά τις συμφωνίες τις οποίες υπογράφουν οι χώρες μέλη με τρίτες χώρες. Δεν θέλουμε να θέσουμε θέματα που έχουν σχέση με την τιμή του αερίου ή με το μέγεθος των ποσοτήτων. Δεν θέλουμε εμείς να θίξουμε την διαπραγματευτική αυτονομία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Οι τιμές δεν μας ενδιαφέρουν. Εμείς μόνο τα διακανονιστικά στοιχεία των συμφωνιών αυτών θα ελέγξουμε γιατί θα μπορούσαν να είναι ασύμβατα με την εσωτερική αγορά. Νομίζω λοιπόν ότι έτσι θα αντιμετωπίσουμε σωστά το θέμα της επικουρικότητας ε, γιατί όπως είπα ε, δεν θα κυκλοφορούν σε καμία περίπτωση ε, πληροφορίες πάνω στις τιμές ή στις ποσότητες υποεμπορία. Ευχαριστώ κύριο Κάραντ αν θέλει να κάνει τι τελικέ παρατηρήσει του. Δεν υποχρεωμένος εάν το θέλει βέβαια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. στην Επιτροπή αυτή βρισκόμαστε όλοι σε παράλληλη πορεία. Στην κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το γεγονός ότι μπορεί μια σύμφωνη όπως το Nord Stream να περάσει από, από τη διακρατική σφαίρα στην ιδιωτική σφαίρα, την εμπορική σφαίρα. Είναι μια ανησυχία θεμητή αυτή, αλλά αυτό που θυμίζει η Κομισιόν είναι ότι η νομοθεσία από την πλευρά της Κομισιόν Σημαίνει απλώ ότι θέλουμε να έχουμε ένα φίλτρο για να βλέπουμε αν αυτέ οι συμφωνίε ευθυγραμμίζονται ή όχι με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αν είναι κάποια σχέδια λοιπόν όπου τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να τα υποβάλουν σε έλεγχο με το να χρησιμοποιούν εμπορικέ συμφωνίε και όχι διακρατικέ ε, συμφωνίε, αυτό είναι ακόμα χειρότερο γιατί αυτό αυξάνει το κίνδυνο για διαδικασία επιπαραβάση και αυξάνει και το κόστος για τις εταιρείες σε τελική ανάλυση το θέμα είναι κατά πόσο αυτές οι συμφωνίες ε, συνάδουν ή, ή όχι με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως δεν είναι τόσο μεγάλος ο κίνδυνος άμα το δούμε έτσι. Και για αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν όταν δίκανε σε αυτή την πρόταση της Κομισιόν πράγματι αντιμετωπίζει μόνο τις νομικές πτυχές των διακρατικών αυτών συμφωνιών. Ξέρουμε όμως ότι στην Πολωνία, και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, της πολωνικής κυβέρνησης που χάρηκε πολύ γιατί συμμετείχε η πολωνική κυβέρνηση σε μια συμφωνία με τη Γιάμαλ και βοήθησε την πολωνική κυβέρνηση. Θα υπάρχουν κυβερνήσεις λοιπόν που θα θέλουν να συμμετέχει η Κομισιόν να τους βοηθήσει και αυτές οι κυβερνήσεις οι οποίες φοβούνται ότι η Κομισιόν θα έρθει να τους βοηθήσει ούτως ή άλλως, εκεί απλώς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι λειτουργεί σωστά το νομικό στοιχείο, ότι υπάρχει η αξιολόγηση από την Κομισιόν για την συμμόρφωση με, τον, ε, με, το, με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εκεί λοιπόν που θέλει κάποιο να έχει την Κομισιόν θα έρθει η Κομισιόν. Εκεί που δεν θέλει θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα δέχονται οι κυβερνήσει το φίλτρο αυτό και την συμμόρφωση με, τον, με τους ευρωπαϊκούς νόμους. Είναι ένα πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια ενιαία στάση στην αγορά ενέργειας. Δεν φτά, μας φτάνει στο στόχο, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα στην σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κλείσει και αυτό το σημείο της τη διάταξη <laughs> και εγώ. Νομίζω ότι φτάνει στις 19-20 του Δεκεμβρίου έχουμε την επόμενη συνεδρίασή μας, αν συμφωνείτε. Μερσή,